Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ που σε αυτή τη δημόσια ακρόαση για, τον, ε, για την νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και την αναθεώρηση των σχετικών οδηγιών και τις ε, μελλοντικέ εξελίξεις που προβλέπονται. Η συνεδρίαση αυτή έχει οργανωθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή ε, Γεωργίας και Ανάπτυξης ΠΕΤΡΟΥ. Θέλουμε να διευκρινίσουμε κάποια από τα άρθρα της οδηγιας 9844 για την προστασία των βιοτεχνολογικών ανακαλύψεων. Τα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διάφοροι εταίροι και το Ευρωκοινοβούλιο έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους σε σχέση με τη δυνατότητα να προβλέψουν ε, προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για ειδικέ ε, λειτουργίες βιολογικές και διαδικασίες βιολογικές, ιδίως μετά από μια απόφαση του Διευρυμένου Συμβουλίου Εφέσεων του Ευρωπαϊκού ε, Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών για το θέμα. Θέλαμε λοιπόν να δούμε τις αρχικές αντιδράσεις του ε, Γραφείου των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζητώντα μαζί με του εκπροσώπου των Επιτροπών Γιούρι και Άγκρη για το μέλλον τη οδηγία βιοτεχνολογικών προϊόντων. Εδώ καλωσορίζω λοιπόν τον συνάδελφο και πρόεδρο τη Επιτροπή Άγκρη, τον κύριο Σικέσκι, και θα του δώσω το λόγο για να κάνει τι ανακτήριε παρατηρήσει του για αυτή την ακρόαση, πρωτού περάσουμε στη σύντομη παρουσίαση τη ε, ε ομιλία τη Επιτροπή. Έχετε τον λόγο. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή ακρόαση, ιδίως τους προσκεκλημένους μας, τους εμπειρογνώμονες. Ελπίζω οι παρουσιάσεις σας να μας διαφωτίσουν σε σχέση με αυτά τα πολύ περίπλοκα ζητήματα. η εκτροφή ε, ειδών, φυτών και ζώων, η καλλιέργεια μάλλον φυτών, είναι ε, ένα θέμα που απασχολεί πάντοτε τους ε, αγρότες και βεβαίως μέσα στα, στις ε, αρμοδιότητες και στα ενδιαφέροντά μας είναι και ο διατροφικός εφοδιασμός, η ασφάλεια του εφοδιασμού Το 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσίασε την γνώμη του για το Ευρωπαϊκό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και για τα βιολογικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Υπάρχει μια σχετική οδηγία όπου γίνεται ε, αναφορά στη δυνατότητα έκδοσης διπλωμάτων ευρωσιτεχνίας σε σχέση με είδη φυτών και ζώων, ότι δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα, ότι πρόκειται για διασταύρωση ή για φυσική επιλογή. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να αποσαφινιστεί πλήρως και να καθοριστούν με σαφήνεια οι εξαιρέσεις. Οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί, οι αγρότες αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα. Γι' αυτό και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία η σημερινή μας συνάντηση ε, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και άλλοι, άλλες πλευρές να μπορέσουν να φωτίσουν διάφορα ζητήματα προκειμένου να διασκεδάσουμε τους φόβους που εκφράζουν οι γεωργοί και οι οργανώσεις τους. Είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο χρειάζεται να συζητηθεί διεξοδικά και με διαφάνεια. Και... Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να περάσουμε τώρα στα αγγλικά, στους προσκεκλισμένους μας. Ο κύριος Γκάλι λοιπόν, ο οποίος είναι δικηγόρος για τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και καταπολέμησης της παραχάραξης από τη Γενική Διεύθυνση Growth, έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά για την Επιτροπή να παρουσιάσει αυτό το έγγραφο της Επιτροπής που εγκρίθηκε πρόσφατα στις 3 Νοεμβρίου. Η Οδηγία 9844 για την προστασία για τις παραχαράξεις είναι ένα μεγάλο επίτευγμα Εάν σκεφτείτε το όλο θέμα και η συζήτησή του ξεκίνησε το 1995 και τελικά η έγκριση ήρθε το 1998. Τότε τα προβλήματα δεν εντοπίζονταν στο βασικό ζήτημα που μας απασχολεί σήμερα, αλλά κυρίως ε, στα φυτά και τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Αυτό που έλεγε η οδηγία για τις βιοτεχνολογικές ε, διαδικασίες είναι αυτά που λέει και το άρθρο 4.1.5 με τα διπλώματα που αποκλείονται και εξαρτούνται τελείως από τέτοιες διαδικασίες. Υπήρξε μία έφεση στο εφετείο από το 2010 η γνωστή υπόθεση ντομάτες και μπρόκολα ένα. και με την ολοκλήρωση της υπόθεσης το συμπέρασμα ήταν ότι δεν μπορεί να υπάρχει δίπλωμα προστασίας, δίπλωμα βεστεχνίας Η τέτοιου είδους ε, διαδικασίες. Η νέα αίτηση υποβλήθηκε στο Γραφείο Τεχνιών, όχι για την ίδια τη διαδικασία, αλλά για το αποτέλεσμα, τα προϊόντα που μπορεί κανείς να παράγει με αυτού του είδους τις διαδικασίες. Η απόφαση του διευρυμένου Προεδρείου του Εφετείου το 2015 για την λεγόμενη υπόθεση ντομάτες μπρόκολα 2 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να υπάρξει δίπλωμα ευρεσιτεχνία για τα προϊόντα τα οποία έχει δημιουργήσει κανεί με αυτού του είδου τι βιοτεχνολογικέ διαδικασίε και υπογραμμίζει η απόφαση ότι αυτό θα ισχύει ακόμη και αν ο μόνος τρόπος να παράξει κανείς ένα τέτοιο προϊόν είναι αυτού του είδους οι συγκεκριμένες βιοτεχνολογικές διαδικασίες. Βεβαίως, η απόφαση αυτή έχει προξενήσει συζήτηση και εδώ στο σώμα σας, στο Ευρωκοινοβούλιο και βλέπετε στη διαφάνεια ότι η Επιτροπή Άγκρη τα συζήτησε αυτά δύση, νομίζω τουλάχιστον ως τώρα ε, Εγώ ήμουν σε μία συνεδρία, αλλά νομίζω ότι συζητήθηκαν τουλάχιστον σε δύο. Υπήρξε ένα ψήφισμα από το Δεκέμβριο του 2015 για το θέμα αυτό. Και πιο πρόσφατα η ομάδα για τα δικαιώματα αυματική ιδιοκτησία, IP και για τα ε, θέματα του copyright, ε, συζήτησε πάλι το θέμα αυτό. Ε, πρόεδρε, να επανέλθω στο ψήφισμα. Ήταν σαφέ, όπω και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι πρέπει να διευκρινιστεί το θέμα που έχει να κάνει με το άρθρο 4 12 παράγραφος 3 και 30 παράγραφος 3 για το ίδιο ζήτημα όλα, την ενδεχόμενη απαγόρευση για την έκδοση διπλώματο ευρεσιτεχνία για προϊόντα τα οποία έχουν προέλθει από συγκεκριμένε βιοτεχνολογικέ διαδικασίε. Η αίτηση αυτή απευθύνθηκε, το αίτημα μάλλον αυτό απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίση η Ολλανδική Προεδρία ανέλαβε το όλο θέμα και οργάνωσε ένα συμπόσιο για το θέμα αυτό. Τα βασικά συμπεράσματα του συμποσίου ήταν μια σειρά από σκέψεις ότι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει ένα σημείωμα με κάποιες ε, ιδέες βασικές για τα θέματα αυτά αλλά και κάποιες προτάσεις περί διαφάνειας, δηλαδή να είναι σαφές ποιο δίπλωμα καλύπτει τι και με τι άλλο μπορεί να, επικαλύπτει, ε, να, να υπάρχει επικάλυψη, ποια δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δηλαδή. Και επίσης το θέμα της πρόσβασης, δηλαδή πώς μπορεί κάποια εταιρεία ή επιχείρηση ή επιμέρους άτομα να έχουν πρόσβαση σε βιοτεχνολογικό υλικό εφόσον θέλουν να περάσουν σε έτοιμα ή νέα προϊόντα. Και επίση τα θέματα τη συνεργασία. Ήταν σαφέ ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Περιστεχνιών και του CPO. Για να βεβαιωθούμε ότι ακολουθούμε τις ίδιες ε, γραμμές όταν αξιολογούμε την ουσία τέτοιου είδου εφευρέσεων ή ανακαλύψεων. Συζητήθηκε επίσης σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις η νομική διάσταση του θέματος στο Συμβούλιο ε, των Υπουργών Γεωργίας και Λίας. αλλά και στο Συμβούλιο ανταγωνιστικότητα το Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο φέτος δηλαδή. Εδώ σίγουρα εκφράστηκαν ανησυχίες από την κοινότητα από την πλευρά των κοινοτρόφων. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αυτό το σημείωμα μόλις στις 3 Νοεμβρίου και το σημαντικό που πρέπει να πούμε εδώ είναι αυτό το σημείωμα δεν είναι νομικό δεσμευτικό. Απλώ δείχνει ποια είναι η γενική αντίληψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την στάση θα που να ακολουθήσουν οι Ευρωπαίοι νομοθέτε, δηλαδή το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, για το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα. Βεβαίω η θέση αυτή δεν δεν προδικάζει το πώ θα τοποθετηθεί εν τέλει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εφόσον εκδικαστεί η υπόθεση <clears throat> εκεί. Το σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλύπτει τρεις πτυχές. Το ζήτημα που ήδη αναφέρθηκε, δηλαδή δυνατότητα προστασίας με δίπλωμα για προϊόντα που ε, έχουν παραχθεί με συγκεκριμένες βιοτεχνολογικές διαδικασίες και το άλλο σκέλος, η ε, πολλαπλή έκδοση αδειών για προστασία δεν καλύπτονται εδώ θέματα τα οποία δεν ζητήθηκε από την Επιτροπή να καλυφθούν. Όπως οι νέε κτηνοτροφικέ ε, τεχνικέ λόγω χάρη, θα ήταν λίγο δύσκολο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερμηνεύσει τα πάντα και να ερμηνεύσει και την πρόθεση του νομοθέτη κυρίω. Επίσης, η περιορισμένη εξαίρεση του κοινοτρόφου δεν συζητιέται, διότι αυτό δεν επίπτει στο πεδίο της οδηγίας 9844. Το πρώτο, λοιπόν, η προστασία από δίπλωμα για συγκεκριμένα προϊόντα που προέρχονται από βιοτεχνολογικές διαδικασίες, η απάντηση της Επιτροπής ήταν να ασχοληθεί με το προπαρασκευαστικό έργο για την οδηγία και να το ξαναμελετήσει. Γι' αυτό το αρχικό άρθρο 4 της πρότασης της Επιτροπής το ξαναείδαμε και είναι σαφές. Εάν διαβάσετε ε, το κείμενο, καταλαβαίνετε ότι τα προϊόντα ή φυτά στα οποία καταλήγουμε με βασικέ τεχνολογικέ διαδικασίε, βιολογικέ μάλλον διαδικασίε, δεν μπορούν να είναι αντικείμενο προστασία από δίπλωμα. Αυτή ήταν η πρώτη πρόταση τη Επιτροπή. Τι έγινε κατά τη διάρκεια τη συζήτηση τώρα. Εσεί στο Κοινοβούλιο είχατε την ιδέα να διαγραφεί το άρθρο αυτό. Δεν σημαίνει όμω αυτό ότι η συγκεκριμένη διαγραφή σημαίνει ότι το Ευρωκοινοβούλιο διαφωνεί με την προσέγγιση μας. Απέναντίας, εάν δείτε την έκθεση που ετοίμασε και συνέταξε ο εισηγητής, ο κ. Ρότλαϊ, αναφέρεται ξεκάθαρα η πρόθεση του Ευρωκοινοβουλίου να μην χορηγήσει ε, διπλώματα ευρεσιτεχνία για συγκεκριμένε βασικέ βιοτεχνολογικέ διαδικασίε, οι οποίε έχουν να κάνουν με διασταύρωση και επιλογή. Και δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτέ τι τεχνικέ. Δεν θα πρέπει να προστατεύονται από δίπλωμα λοιπόν αυτέ, αλλά ούτε και τα προϊόντα που αποκτώνται από τέτοιου είδου ε, διαδικασίε. Ήταν ε, σαφέ λοιπόν αυτό στην έκθεση του κ. Ρότλεϊ. Δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση από το Κοινοβούλιο να ακολουθήσει αυτή την άγουσα. Τι έγινε μετά. Η Επιτροπή μελέτησε και τις τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο, ιδίως για τα φυτά. Τις ενέκρινε και το Συμβούλιο και καταλήξαμε στο νέο άρθρο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Νέο άρθρο που αντί να αναφέρεται μόνο στα φυτά και τα ζώα, αναφέρεται μόνο στο βιολογικό υλικό. Τι λέει το άρθρο αυτό το 3 εν ώψη των προπαρασκευαστικών εργασιών είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι υπάρχουν δύο δυνατότητες όπου μπορεί να λάβει κανείς δίπλωμα όταν το ε, βιολογικό περιεχόμενο, το βιολογικό υλικό δεν έχει σχέση με το περιβάλλον του, όταν είναι αποτέλεσμα μια διαδικασία, μια επεξεργασίας δηλαδή. Ε, και δεύτερον, όταν υπάρχει μια τεχνική επεξεργασία για να παραχθεί το προϊόν, τότε Μπορούμε να θεωρήσουμε την τεχνική διαδικασία και βιολογική ενδεχομένω. Άρα το συμπέρασμα για το άρθρο αυτό είναι ότι δεν μπορεί να πάρει κανεί δίπλωμα για τα προϊόντα που αποκτώνται από βασικέ βιολογικέ διαδικασίε. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε. Αν δείτε λίγο το σημείωμα, το κείμενο είναι στη σελίδα 7, όπου η Επιτροπή δηλώνει ότι η πρόθεση του νομοθέτη ήταν σαφώς να αποκλείσει την προστασία των προϊόντων αυτών από δίπλωμα και τώρα μιλάμε μόνο για φυτά. Αλλά η ίδια λογική μπορεί να εφαρμοστεί και στα ζώα. Δεν μπορεί κανείς να πάρει δίπλωμα για την προστασία ζώου το οποίο έχει ε, δημιουργηθεί από βιολογικές διαδικασίες που μπορούν να, να θεωρηθούν ουσιαστικές. Τα άλλα δύο συμπεράσματα, επειδή δεν υπάρχει και χρόνο και δεν είναι και το βασικό θέμα που πρέπει να συζητήσετε σήμερα το απόγευμα, είναι ότι θυμηθείτε στο σημείωμα ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί την ε, στάση για την πολλαπλή προστασία από άδειε, την πολλαπλή έκδοση αδειών μάλλον και το σχετικό άρθρο. Εκεί διευκρινίζει τη στάση τη Επιτροπή. Και το τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με την πρόσβαση σε βιολογικό υλικό και την πρόσβαση στα δείγματα τα οποία τηρεί ο οργανισμός στον οποίο έχει ε, να αποτεθεί ευθύνη να προστατεύει το βιολογικό αυτό υλικό. Αυτό θα το μελετήσει περαιτέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας έχει αποστείλει το σχετικό σημείωμα. Θα δούμε τα... το υπόμνημά της δηλαδή, θα δούμε τα επόμενα βήματα. Πάντω, νομίζω πρώτο βήμα είναι η διοργάνωση αυτή τη ίδια τη ακρόαση. Σα ευχαριστώ λοιπόν που οργανώσατε τη συζήτηση αυτή για το υπόμνημα και ελπίζω να τα συζητήσουμε και σε επίπεδο Επιτροπή και βεβαίω είναι δικό σα το θέμα να αποφασίσετε τι ε, συνέχεια πρέπει να δοθεί σε αυτό το υπόμνημα. Στο επίπεδο του Συμβουλίου νομίζω είναι σημαντικό να πούμε ότι χθες μόλις έγινε συζήτηση για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας από τα διάφορα και εκεί το Συμβούλιο έλαβε γνώση του, του υπομνήματος, του σημειώματος και κάποιες χώρες, ιδίως οι κατοχώρες και η Αυστρία, ε, συμφώνησαν μάλιστα και τάχθησαν υπέρ των συμπερασμάτων του υπομνήματος. Τώρα η ομάδα IP Επιτροπή συνεδριάζει στι 16 Δεκεμβρίου. Τότε είναι προγραμματισμένη η επόμενη συνάντηση για να συζητηθεί αυτό το υπόμνημα τη Επιτροπή, ενδεχομένω με, την, με τον το επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλίας στα μέσα του επόμενου μήνα να ασχοληθεί με το θέμα. Μπορεί και αυτό και πάλι να ε, εξεταστεί από τα διάφορα. Εκεί μπορεί να υπάρξει κάποιο σχολιασμό από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα επίση τον ε, Φεβρουάριο. Και να πω ότι σημαντικό είναι το επόμενο να συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί θα υπάρξουν επιπτώσεις για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Έλα κυρία Φρόιλιγκερ, η επόμενη μιλήτρια θα μα τα πει καλύτερα όλα αυτά. Να σα πω απλώ ότι την περασμένη εβδομάδα, τη Δευτέρα συζητήθηκαν αυτά στην Επιτροπή Νομοθεσία για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνία. και περιμένουμε να συνεχιστεί η συζήτηση και σε επίπεδο οργανισμών διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία και του χρόνου. Η κυρία Φρόιλιγκερ λοιπόν θα μα τα εξηγήσει καλύτερα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank Ευχαριστώ πολύ, δόκτωρα Γκάλ. Και θα ήθελα να καλέσω την κυρία Μάργκοτ Φρούλιγκερ, κυρία Διευθύντρια για του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων ε- Ευρεσιτεχνίας, για θέματα νομικά και πολυμερή. Έχετε 10 λεπτά. Thank you, Madam Chair, and... Uh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Μου ζητήθηκε να σας παρουσιάσω το νομικό πλαίσιο βάσει του ΕΠΙΟΥ, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας εξετάζει και χορηγεί διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τα φυτά. Πριν ξεκινήσω την παρουσίασή μου θα ήθελα να τονίσω ότι το γραφείο μας είναι μια τεχνική οργάνωση. Δεν έχουμε πολιτική ε, κλίση. Εφαρμόζουμε το νόμο ως έχει. Και αυτή η υποσημείωση είναι εξαιρετικά σημαντική και γι' αυτό με αυτή την ειδοποίηση ε, ξεκινήσαμε τη διαδικασία διαβούλευσης με τα μέλη μας. Τα περισσότερα είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε το θέμα εκ του σύναγκης εάν τα συμβαλόμενα κράτη-μέλη, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας το ζητήσουν. Επομένως, νομικό πλαίσιο για βιοτεχνολογικές εφευρέσεις και επινοήσεις. Διέπεται καταρχάς από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Εύρεση Τεχνίας που, επικυρια... που προηγείται της σχετικής οδηγίας. Το ευρωπαϊκό, η σύμβαση αυτή ερμηνεύεται από το Συμβούλιο Προσφυγών ή Εφέσεων που έχουμε, το οποίο είναι ανεξάρτητο και είναι σημαντικό να κατανοήσει κανείς ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δεν έχουμε καμία επιρροή πάνω στην ομολογία του Συμβουλίου ε, Προσφυγών. Έχουμε την οδηγία που βλέπετε στην οθόνη που έχει εφαρμοστεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Θα έρθω ξανά στην οδηγία και έχουμε και την εθνική νομοθεσία από τη στιγμή που τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας μπορούν να τεθούν σε ισχύ αλλά και να αμφισβητηθούν και να γίνουν αντικείμενο ανάκλησης ενώπιον εθνικών δικαστηρίων. Η οδηγία λοιπόν αυτή έχει εφαρμοστεί με ε, τους εφαρμοστικούς κανονισμούς ε, του 99. Και αυτός ο τρόπος εφαρμογής επιλέγει για να αποφευχθεί αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα διπλώματα τεχνίας. Μία διαδικασία αναθεώρησης η οποία θα ήταν εξαιρετικά μακροχρόνια και περίπλοκη. Και γι' αυτό διαλέξαμε να εφαρμόσουμε την οδηγία μέσα από εφαρμοστικούς κανόνες αναπερίπτωση. Δηλαδή κάθε άρθρο της οδηγίας, π.χ. βιοτεχνολογία, βιολογικές ε, ε, εφευρέσεις, έχει αντικατοπτριστεί και εφαρμοστεί με αντίστοιχο εφαρμοστικό κανόνα. Και αυτοί οι εφαρμοστικοί κανόνες αποτελούν επιπρόσθετο τρόπο ερμηνείας των κανονισμών και κανόνων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας αυτή καθε αυτή. Και παρόλο που το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας είναι εκτός νομικής τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνήθως το γραφείο μας και το Συμβούλιο Προσφυγών ακολουθεί την ερμηνεία της οδηγίας όπως αυτή αναφέρεται στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και αυτό έχει συμβεί στην περιβόητη υπόθεση Κέσλερ με τα βλαστοκύτταρα όπου υιοθετήσαμε και εφαρμόσαμε νομολογία που συνάδει απολύτως με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ποια είναι η τρέχουσα πρακτική και πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τα φύτα. Υπάρχει αποκλεισμός δεν μπορεί να έχει κανείς διπλώματα ευρεσιτεχνίας για ε, φυτά και ποικιλίε αυτά καθεαυτά και αυτές καθεαυτές. Βιολογικές διεργασίες για την παραγωγή φυτών αποκλείονται σαφέστατα βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ε, Διπλωμάτων Βροσιτεχνίας και της Οδηγίας για την Βιοτεχνολογία. Ως εκ τούτου δεν δίνονται διπλώματα για τέτοιου είδους διεργασίες. Άρα το ζήτημα που είναι αφιλεγόμενο, που ε, έδωσε λόγο σε πολλές αντιδράσεις και που διευκρινίστηκε είναι το εξής. Το γεγονός ότι μπορούν να δοθούν διπλώματα χνές για προϊόντα που προκύπτουν από άμεσες βιολογικές διαδικασίες είναι πρόβλημα και αυτά τα διπλώματα έχουν, ε, ε, αυτά τα θέματα έχουν ενταχθεί στην ε, συζήτηση για την ομολογία για τις υποθέσεις της ντομάτας και του μπρόκολου 2. Γιατί εκεί το Συμβούλιο Προσφυγών βρήκε ότι δεν μπορούν να δοθούν διπλωματεύρεση τεχνίας στις διεργασίες, ότι δεν υπάρχει αποκλεισμό από τα φυτά, από τα διπλώματα τεχνίας για τα φυτά, ακόμα και αν έχουν προκύψει από βιολογικές διεργασίες. Είναι πολύ τεχνικές εξηγήσεις και θα τις παρακάμψω γιατί μου ζητήθηκε να είμαι εξαιρετικά σύντομος και για να δώσω περισσότερο χώρο στη συζήτηση. Έχουμε παρακολουθήσει τις αποφάσεις ντομάτα 2 και μπροκόλο 2 ε, στο Συμβούλιο Προσφυγών. Ξεκίνησε μία συζήτηση με τα συμβαλόμενα κράτη-μέρη ε, στην αντίστοιχη επιτροπή και ζητήσαμε την άποψη των συμβαλόμενων κρατών για αυτή την ομολογία, την πρόσφατη του Συμβουλίου των Προσφυγών. Και ο πρόεδρος της Επιτροπής για το Δίκαιο των Διπλωμάτων Ευρεσιταχνίας μετά τις συζητήσεις αυτές του, του Μαΐου του περασμένου κατέληξε σε απόφαση η οποία συνοψίζεται ως εξή. Η κατάσταση στα συμβαλόμενα κράτη ε, συνοψίζεται σε τρεις κατηγορίες. Πρώτον, η πρώτη ομάδα συμβαλόμενων κρατών είναι αυτή όπου το εθνικό δίκαιο και η εθνική πρακτική κατά συνέπεια συνάδει με τη δική μας νομολογία του Συμβουλίου ε, Προσφυγών. Υπάρχει μια δεύτερη ομάδα χωρών και σημαντική όπου το Εθνικό Δίκαιο διαφέρει από την ερμηνεία που έχει δώσει στο θέματα αυτά το Συμβούλιο Προσφυγών και αυτά τα κρατημέλη έχουν εκφράσει ισχυρές ανησυχίες για την ομολογία του Συμβουλίου Προσφυγών. Και στη συνέχεια υπάρχει μια τρίτη κατηγορία χωρών όπου η κατάσταση δεν είναι απολύτως σαφής. Έχουμε συνεχίσει τη συζήτηση με τα κρατημέλη στις 21 Νοεμβρίου του 2016 μετά το σημείωμα την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάστηκε εδώ σήμερα. Και το αποτέλεσμα αυτό ήταν ε, ενδιαφέρον. Δηλαδή, αρκετά συμβαλόμενα κράτη τάχθηκαν ξεκάθαρα υπέρ του σημειώματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από αυτό το μεγάλο αριθμό κρατών μελών που είναι υπέρ της ερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε και έναν άλλο αριθμό σημαντικό ε, συμβαλόμενων κρατών που θα ήταν υπέρ της αλλαγής του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα διπλώματα ευρωσιτεχνίας και που θα ήταν υπέρ της τροποποίησης και προσαρμογής των εφαρμοστικών μας κανόνων έτσι ώστε οι κανόνες αυτοί να ευθυγραμμιστούν με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. και ορισμένες αντιπροσωπείες είπαν ότι δεν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, ότι η απόφαση θα ήταν πρόημη και ότι πρέπει να περιμένουμε για την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν αυτό το δικαστήριο επιβεβαιώσει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τότε και μόνο τότε θα πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Επομένως, με, τη βάση, με βάση όλες αυτές τις συζητήσεις, η Επιτροπή σημειώνει ότι εμείς συνεχίζουμε τις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη, ότι Προετοιθέμεθα να παρουσιάσουμε στα συμβαλόμενα κράτη μας ένα έγγραφο το οποίο θα σκεγγραφεί τις αποκλίνουσες μεταξύ τους επιλογές και μία από αυτές τις επιλογές θα είναι και η τροποποίηση του νομικού μας πλαισίου μέσω της έλευσης τροποποιήσεων στους εφαρμοστικούς κανόνες. Και οφείλω να τονίσω για άλλη φορά το γεγονός ότι από τη στιγμή που είμαστε τεχνική οργάνωση και εφαρμόζουμε τον νόμο, μόνο προτάσεις μπορούμε να υποβάλλουμε, τις, οι οποίες για να ισχύσουν πρέπει να υιοθετηθούν και να εγκριθούν από τα συμβαλόμενα κράτη-μέλη μας. Εν όψη λοιπόν και με βάση την, το σημείωμα και την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώσαμε αποφασίσαμε να ε, αναστείλουμε την έκδοση αποφάσεων για όλους αυτούς τους φακέλους και για όλα αυτά τα θέματα, για φυτά δηλαδή που προκύπτουν από κατ' ουσίαν βιολογικές διεργασίες. Επομένως, εκκρεμεί η έκβαση της συζήτησης με τα κράτη-μέλη για το κατά πόσο θα πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο ή όχι. Ήδη προσπαθούμε η πρακτική των εξεταστών μας να ευθυγραμμιστεί με το, την ανακοίνωση, το σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τα θέματα της ποικιλία των, των φυτών μπορώ να τα παρακάμψω. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ κυρία Φρύλιγκερ για την παρέμβασή σας. Έχουμε τώρα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, ερωτήσεις, να δώσετε απαντήσεις, να γίνουν σχόλια αξιοποιούμε την παρουσία των καλεσμένων μας. Η κυρία Χόιμπους. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη γιατί πρέπει να φύγω, γιατί έχω μια ψηφοφορία αλλού. Παρ' όλα αυτά θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Αυτό που μου λείπει είναι μια ισχυρή φωνή για τους αγρότες και τις αγρότες, ε, αγρότησες, για τα συστήματα τροφοδοσίας, γιατί αν θέλουμε να διατηρήσουμε την πρόσβαση των γεωργών στους σπόρους, πρέπει να εξασφαλιστεί και αυτό. Δηλαδή, το να, ε, να αποκατασταθεί η δυνατότητα των γεωργών να ανανεώνουν τους σπόρους τους και να τους αντικαθιστούν ή να τους ανταλλάσσουν. Και αυτό ε, έχω καταλάβει ότι η Κομισιόν θέλει να απαγορεύσει και να κατακαιρματίσει το σύστημα του Safe Seed. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι όλα όσα κάνουμε στην εκτροφή είναι, βασίζεται σε όσα έκαναν επί χιλιάδες χρόνια οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες οι οποίοι ποτέ δεν αποζημιώθηκαν για οτιδήποτε από, από όλα αυτά που έκαναν και τώρα ξαφνικά ε, δεσμεύεται ε, μια διεργασία ως πνευματική ιδιοκτησία αλλά ε, για μένα αυτό που είναι σημαντικό είναι να μην κινδυνεύσει η δυνατότητα των γεωργών να εκτρέφουν, να ανανεώνουν και να επαναχρησιμοποιούν τους σπόρους τους. Γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κάποιες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που ήδη ε, κατέχουν το 70 90% του μεριδίου αγοράς των σπόρων να φροντίσουν αυτοί και μόνο για το μέλλον μας. Αντιθέτως, πρέπει να ε, εμπιστευτούμε την τύχη του μέλλοντος της γεωργίας στους γεωργούς γιατί αλλιώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητούμε ε, και για ζητήματα όπως είναι η βιοπικιλότητα γιατί και αυτό το θέμα συνδέεται με αυτό που συζητούμε σήμερα. Ευχαριστώ και πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ. Επόμενος ε, ομιλητής είναι ο κύριος Χούτεμαν. Ευχαριστώ πολύ ε, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Βρουσιτεχνιών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω ένα ερώτημα προς το γραφείο. Τονίσατε ήδη τη συνέχεια που έχει δοθεί. Υπάρχουν κάποια συμβαλόμενα κράτη που θέλουν πράγματι να αλλάξουν το περιεχόμενο των εφαρμοστικών κανόνων. Εγώ ελπίζω πραγματικά να το καταφέρουν. Ε, νομίζω ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ήταν σαφέστατο και έτυχε πολύ μεγάλης πλειοψηφίας. Ωστόσο το ερώτημά μου είναι, αν θα αλλάξετε τους εφαρμοστικούς κανόνες, αρκεί αυτό, δεν θα δίνονται δηλαδή διπλώματα έβρεση τεχνίας από την πίσω πόρτα για παράδειγμα. Μπορείτε να το εγγυηθείτε αυτό. Και μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παραγράφους 8-9 του άρθρου του, της ε, ε, οδηγίας για τα βιοτεχνολογικά προϊόντα. Θα υπάρχει δυνατότητα χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε προϊόντα που έχουν προκύψει από βιοτεχνολογικές ε, διεργασίες. Επίσης, ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να δημοσιεύσει έκθεση για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του δικαίου περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, όπως αναφέρεται ε, μέσα στο κείμενο της ε, οδηγία, της προτινόμενης οδηγίας, γιατί για το γνώμη μου κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβεί. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άγνου. Thank you. I think I've... Ευχαριστώ πολύ. Κάτι έμαθα και σήμερα. Ε, για τον πρώτο ομιλητή μου άρεσαν πολύ αυτές οι, οι νέες προφορίες για την εκτροφή ζώων και φυτών είπατε ότι υπάρχουν, δύο, υπάρχουν νέα στοιχεία. Ότι θα πρέπει καταρχάς να, ε, να συμψηφιστούν με, του, με τα γενετικά τροποποιημένα και να απαγορευτούν. Είπατε επίσης ότι υπάρχουν διαφορές από την άλλη πλευρά μεταξύ των, ε, της ε, καλλιέργειας φυτών και των γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών γιατί είπατε ότι με βάση τις νέες διαδικασίες που υπάρχουν μπορούν να επιτευχθούν και προϊόντα με φυσικές, με φυσιολογικές διεργασίες γι' αυτό θα πρέπει να είναι εντελώς ξεχωριστό ε, κομμάτι τα μεταλλαγμένα. Επίσης, το τρίτο, είπατε ότι ε, όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την καλλιέργεια, την άρδευση, αφορούν και σχετίζονται με την ε, ε, εκτροφή φυτών και ίσως θα μπορούσατε να, να μου δώσετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Για τη δεύτερη ομιλήτρια θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Η ζωή, δε, οι μορφές ζωής δεν, δεν μπορούν να, να ε, πατενταριστούν. Ωστόσο, ένα προϊόν, ένα ζυμαρικό, για παράδειγμα, το οποίο βασίζεται σε ένα είδος φυτού, μπορεί να πατενταριστεί. Το κατάλαβα σωστά. Ωραία, ευχαριστώ. Έχουμε 10 λεπτά για να ακούσουμε τις απαντήσεις των προσκεκλημένων μας και μετά θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτού του θέματος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω στις διάφορες ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στην Επιτροπή. Όλες εάν τα καταφέρω και αν μου ξεφύγει κάτι, από τώρα ζητώ συγγνώμη. Για το αν θα ήταν δυνατό να κοιτάξουμε τα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας για να καταλήξουμε στο ίδιο αποτέλεσμα, προστασία με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η απάντηση είναι σαφής. Όχι. Όχι, δείτε το κεφάλαιο αυτό έχει να κάνει με την προστασία και όχι με τα διπλώματα αυτά καθεαυτά. Για το θέμα του πώς θα χρησιμοποιούνται τα διπλώματα, όλα αυτά υπάρχουν και διθετώνται στο πρώτο άρθρο. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό πίσω πόρτα ως παραθυράκι για να λύσουμε άλλα ζητήματα για τις βιολογικές διαδικασίες και για το άρθρο 16C, 16Γ που αναφέρατε, το σημειώνω. Όμως να ενημερώσω ότι η Επιτροπή, αν και το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο θα αποφασίσουν ε, τι θα κάνουν ε, με τη βούλησή τους ως νομοθετών, ε, κατά πόσον η απόφαση της Επιτροπής είναι σωστή. Εμείς καταγράφουμε τη δική σας άποψη και αυτό βεβαίως σχετίζεται και με το ερώτημα που τέθηκε για τις νέες κτηνοτροφικές μεθόδους. Είναι ένα θέμα που μπορεί να καλυφθεί από την έκθεση αυτή, διότι είναι πραγματικά ένα ερώτημα αρκετά ολιστηρό Ε, είναι ένα θέμα λοιπόν εδώ που μπορεί να προκαλέσει διαφορετικές αντιδράσεις ε, σε μια τέτοια είδους έκθεση και είναι δύσκολο να προδικάσει κανείς αν μιλάμε για γενετικό τροποποιημένο οργανισμό ή ένα συμβατικό προϊόν. Η μόνη δυνατότητα της Επιτροπής θα ήταν να διευκρινίσει το καθεστώς της έκτασης του διπλώματος για τέτοιες διαδικασίες ή όχι αλλά δεν θα λάβουμε θέση για τον χαρακτηρισμό αυτών των προϊόντων με αφορμή τη συγκεκριμένη έκθεση ή οδηγία. Και μετά για τον πρώτο ίσως ομιλητή, μια αναφορά στα δικαιώματα των γεωργών κτηνοτρόφων, διότι και το άρθρο 11 με το περιεχόμενό του είναι σημαντικό, πρέπει να το γνωρίζουν τα μέλη της Επιτροπής αυτής, για τα δικαιώματα των γεωργών και εκτινοτρόφων να χρησιμοποιούν το 6 και τα προϊόντα αυτά. Υπάρχουν κάποιες ε, εγγυήσει, κάποια χέγγια που παρέχει η οδηγία. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλα τα απάντησα. Τουλάχιστον αυτά που απευθύνονταν σε μένα. Να, να δώσω το λόγο στην κυρία Φρόλιγκερ. I ναι, μου ζητήθηκε να απαντήσω στα ερωτήματα που απευθύνθηκαν και στον πρόσωπο της Επιτροπή. Ότι ακόμη και με την αλλαγή των εφαρμοστικών κανόνων θα εξαιρούσαμε την δυνατότητα έκδοσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για προϊόντα που έχουν προκύψει από βιολογικές διεργασίες και αν αυτό θα αρκούσε γιατί δεν θα υπάρχει κάποια πίσω πόρτα. Αυτό που μπορώ να επαναλάβω είναι η απάντηση που έχει δοθεί ήδη από, την, ε, από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Η οδηγία διαρθρώνεται σε διάφορα τμήματα και καθώς η δυνατότητα χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ρυθμίζεται στο κεφάλαιο 1, στο κεφάλαιο 2 Εκεί δεν ρυθμίζεται το ζήτημα της δυνατότητας έκδοσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Είναι δε πρακτική του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας να εκδίδει σαφείς κατευθυντήρες γραμμές για τους ελεγκτές μας. Αν στο μέλλον αλλάξουμε το εκτελεστικό εφαρμοστικό πλαίσιο, τότε σίγουρα θα προβλέπεται μια τέτοια εξαίρεση για προϊόντα που έχουν προκύψει από βιολογικές διεργασίες. Δεν θέλουμε να δίνονται διπλώματα ευρεσιτεχνής ε, σε φυτά ε, από την πίσω πόρτα γιατί αυτό δεν θα ήταν ούτε καν προς το συμφέρον των ετούντων. Θα δημιουργούσε απλώς νομική αβεβαιότητα γιατί αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μπορούν θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενα δικαστικών διαμαχών στα εθνικά δικαστήρια κτλ. κτλ. Όσον αφορά το όριο μεταξύ της ε, προστασίας των ποικιλιών φυτών και της δυνατότητας έκδοσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ο αποκλεισμός από την έκδοση ε, διπλωμάτων για ποικιλίε φυτών Ε, δομείται, ε, ε, έχει, μια πολύ στενή, ένα πολύ στενό περιθώριο ερμηνείας. Αφορά τις ποικιλίε φυτών, ιστόσο υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις όπου υπάρχουν εφευρέσεις βιοτεχνολογικές οι οποίες έχουν ε, συμπεριλάβει ενδεχομένως και κάποια φυτά, χωρίς ωστόσο να, έχει, να έχουν καταλήξει ε, ως τελικό προϊόν σε ένα νέο φυτό. Εκεί επιτρέπεται η έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε αυτές τις περιπτώσεις. Ε, Κυρία Φρόλιγκερ, τελειώσατε. Αυτά, ωραία. Ε, συγγνώμη, ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. τον κύριο Ραν Γκάλ και την κυρία Μάργκοτ Φρόλιγκερ που ήταν η προσκεκλημένοι μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Θα ξανασυζητήσουμε το ζήτημα αυτό και στο μέλλον και περνάμε στο επόμενο θέμα της σημερινής σας διάταξής μας. Συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο σημείο. Στο σημείο 32, Είμαι συγκήτρια για την ε, σύνταξη της γνωμοδότησης όσον αφορά το geoblocking, του γεωγραφικού αποκλεισμού και θα μιλήσω πολωνικά. Βάλτε σας παρακαλώ τα ακουστικά σας. Και θα ήθελα, παρακαλώ, να κάνετε λίγη ησυχία. Ε, λοιπόν, η γνωμοδότησή μου αφορά τον κανονισμό που έχει ως θέμα του τον γεωγραφικό αποκλεισμό Η στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά περιλαμβάνει και νέους κανόνες για να καταπολεμηθεί το, το ανέτιο, ε, ο ανέτιος γεωγραφικός αποκλεισμός καθώς και άλλες μορφές διακρίσεις που οφείλονται στον τόπο κατοικίας, στον τόπο εγκατάστασης ή της οικονομικής δραστηριότητας. Μιλούμε για την καπιτολέμηση ε, διακρίσεων ε, στην πρόσβαση μόνο και μόνο επειδή βρίσκεται κανείς στο ένα ή στο άλλο κράτος μέλος. Ο κανονισμός λοιπόν για τον γεωγραφικό αποκλεισμό ε, επιδιώκει διάφορους ε, σκοπούς ε, μεταξύ αυτών είναι η υποστήριξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών. Ε, καταναλωτές σκοπός είναι να έχουν καλύτερη και πιο εύκολη πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Ταυτόχρονα όμως οι πάροχοι οφείλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους διασυνοριακά. Γιατί δεν επιτρέπεται να ε, κάνουν διακρίσεις εις βάρος πελατών από άλλες μέλη. Οι αρχέ αυτές είναι καλές και τις συμμερίζομαι. Ωστόσο πρέπει ε, να βελτιώσουμε την πρόταση κανονισμού προκειμένου να μπορούν πράγματι να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω δύο ε, οπτικές. Αφενός την οπτική του καταναλωτή. Ο μέσος καταναλωτής πολλές φορές ή πολύ πιθανόν να μην γνωρίζει καν τι, τι σημαίνει ο όρος γεωγραφικός αποκλεισμός ή μπορεί να θεωρεί ότι αφορά το γεγονός ότι δεν μπορεί για παράδειγμα να δει ένα, ένα ποδοσφαιρικό αγώνα επειδή βρίσκεται σε άλλη χώρα. Πολύ πρόσφατα ο κύριος Άγνους είπε ότι εδώ στις Βρυξέλλες δεν μπορεί να παρακολουθήσει τους εστονικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες στη τηλεόραση. Λόγω αυτής της τοποθέτησης, αυτής της δήλωσης, είχαμε θεωρήσει ότι ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να αναλάβει δράση προκειμένου ο καθένας να μπορεί να δει ό,τι θέλει στη χώρα του. Μιλώ για δωρεάν ε, υλικό όταν βρισκόμαστε στην ε, χώρα καταγωγής μας, στην πατρίδα μας. Τελικά όμως τα πράγματα μάλλον δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ε, θα συνεχίσουμε να μην έχουμε πρόσβαση σε αυτό το υλικό ε, όταν βρισκόμαστε σε άλλη χώρα. Διότι η μεταρρύθμιση που προτείνεται δεν αφορά τον γεωγραφικό αποκλεισμό. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει τον πλήρη αποκλεισμό αυτών, αυτού του ψηφιακού περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Καταλάβατε αυτό που, που, σας, ε, που σας είπα, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ σαφές. Εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω γιατί οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες και οι άλλες υπηρεσίες που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ήταν το βασικό και ε, ουσιαστικό αντικείμενο του γεωγραφικού αποκλεισμού αποκλείονται τελικά από την πρόταση που υπευλήθη. Γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω μια τροποποίηση του άρθρου 4 θα πρότεινα εδώ να μην γίνεται λόγος για οπτικοακουστικές υπηρεσίες, αλλά ε, για ηλεκτρονικά βιβλία, e-books, για παιχνίδια, για μουσική, δηλαδή λογισμικό, μουσική, βιβλία και παιχνίδια υπολογιστή. Και θέλω πραγματικά να το σκεφτούμε πώς θα μπορούσαμε να λύσουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αυτό το πρόβλημα του γεωγραφικού αποκλεισμού. Θεωρώ ότι πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ώστε να συμπεριλαμβάνει και τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όταν ο πάροχος αυτός ε, κατέχει αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα ξανακούσουμε παράπονα όπως αυτά που ακούμε πολύ συχνά, ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε υλικό στο οποίο δικαιούμαστε κανονικά πρόσβαση όταν βρισκόμαστε στην πατρίδα μας. Θέλω να το σκεφτούμε. Αν θεωρείτε ότι στο άρθρο 4 για οποιονδήποτε λόγο. Δεν θα καταφέρουμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση, αν και πιστεύω ότι όλοι μας είμαστε πρόθυμοι να βρούμε κάποιον συμβασμό, θα μπορούσαμε στο άρθρο 9, σημείο 2, να ε, αναφέρουμε ρητός αυτές τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει στο μέλλον κατά τη γνώμη μου, να είναι υποχρεωμένη να επανέλθει στο, στο θέμα αυτό, ίσως στο πλαίσιο κάποιας αναθεώρησης. Ξέρω ότι το θέμα αυτό είναι αμφιλεγόμενο, αλλά ε, ε, η γνώμη μου είναι ότι αυτή, αυτό θα πρέπει να είναι το, ε, ο, η μελλοντική μορφή του γεωγραφικού αποκλεισμού. Δηλαδή να έχουμε πρόσβαση όπου και αν βρισκόμαστε. Τώρα θέλω να δούμε και το θέμα από τη σκοπιά του παρόχου. Από τη σκοπιά του παρόχου το σημαντικότερο είναι το ισχύον δίκαιο όσον αφορά τις συμβάσεις του με, τον καταναλωτή. Πρόκειται για το δίκαιο, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι ε, εκεί όπου εδρεύει ο πάροχος ή το δίκαιο της χώρας όπου εδρεύει ο καταναλωτής. Ο ε, οι πάροχοι δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να είναι εξοικειωμένοι με 24 διαφορετικά νομικά συστήματα. Ο κανονισμός λέει ξεκάθαρα ότι ε, στις συμβάσεις αυτές ισχύει το δίκαιο του, της χώρας στην οποία εδρεύει ο καταναλωτής. Σωστό, όμως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο γεωγραφικός αποκλεισμός αποτελεί έναν περιορισμό της οικονομικής ελευθερίας του παρόχου, διότι ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να μην κάνει διακρίσεις εις βάρος των αλλοδαπών καταναλωτών. Αυτό σημαίνει ότι ο πάροχος ε, ενδέχεται να έχει μια οικονομική δραστηριότητα σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, έχει δεχτεί, για παράδειγμα, τη στοιχεία της πιστοτικής κάρτας ε, από κάποια άλλη χώρα, ε, ακόμη και αν ο πελάτης του έχει την έδρα του, τη μόνιμη κατοικία του σε άλλο κράτος. Ωστόσο, ο πάροχος δεν έχει υποχρέωση να παραδώσει τα προϊόντα σε μια άλλη χώρα. Ας σκεφτούμε λιγάκι πώς θα δημορφωθεί η κατάσταση ένας πελάτης ε, διαμένει μόνιμα εκτός Ισπανίας, για παράδειγμα, αλλά του αρέσει πάρα πολύ μια πολύ ε, γνωστή ισπανική μάρκα και στο, στο, στην ιστοσελίδα αυτής της ισπανικής ε, μάρκας μπορεί να αγοράσει ε, πολύ φθηνά τα προϊόντα αυτά από ότι στην ίδια του τη χώρα σε ένα κατάστημα. Λοιπόν, μένει στην Πολωνία, ε, θέλω να αγοράσω ε, ρούχα σε αυτή την ισπανική ιστοσελίδα μέσω του ίντερνετ, με την πιστοτική μου κάρτα κτλ. κτλ. Σήμερα δεν μπορώ να το κάνω αυτό, στο μέλλον όμως θα μπορώ να το κάνω αυτό και θα πρέπει να επιλέξω εγώ, να αποφασίσω εγώ αν θα κάνω τις αγορές μου στην πολωνική ε, ιστοσελίδα ή στην ισπανική ιστοσελίδα. Ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει. Βέβαια, ανακύπτουν και ορισμένα ζητήματα σε σχέση με τι επιστροφέ. Αν δηλαδή το, το προϊόν είναι ελαττωματικό, θα πρέπει να το επιστρέψει στην Ισπανία ή στην Πολωνία. Ο πελάτης λοιπόν θα πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τα νομικά συστήματα της Ισπανίας και της Πολωνίας ή θα πρέπει απλά να μπορεί να κάνει την επιλογή. Φυσικά και δεν έχει ε, υποχρέωση να, ε, ε, δεν έχει υποχρέωση να πραγματοποιήσει τις αγορές του στην Ισπανική ιστοσελίδα και ως εκ τούτου φυσικά δεν έχει και καμία υποχρέωση να γνωρίζει το, το Ισπανικό νομικό σύστημα. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι μήπως τελικά η κατάργηση του γεωγραφικού αποκλεισμού δημιουργήσει προβλήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί ακριβώς θα τις αναγκάσει να είναι εξοικειωμένε και να γνωρίζουν τα νομικά συστήματα όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα είναι προφανές, καμία μικρομεσαία επιχείρηση δεν μπορεί να συντηρήσει νομικό τμήμα το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το καθήκον. Παρ' όλα αυτά θέλουμε όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να πολλούν τα προϊόντα τους σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε έναν καλό κανονισμό. Χρειαζόμαστε νομική ασφάλεια για τους παρόχους, οι οποίοι δεν θα πρέπει να παραβιάζουν τον νόμο. Ταυτόχρονα θα πρέπει ωστόσο να προστατευτούν και οι καταναλωτές. Είναι δύσκολο το έργο αυτό να συνδυαστούν και τα δύο αυτά καθήκοντα, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Και πρέπει να, το σκεφτούμε, να σκεφτούμε τι μορφή θα έχει αυτό το πράγμα στην πράξη, στο μέλλον πόσο μεγάλε είναι για παράδειγμα οι διαφορέ μεταξύ των καταναλωτών στι διάφορε χώρε μπορεί και, και οι διατάξει οι ισχύουσες. Ε, σε κάποιε χώρε μπορεί να υπάρχει διαφορά όσον αφορά την περίοδο εγγύηση που παρέχεται. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι αυτά ε, είναι δευτερεύοντα ζητήματα τα οποία με κάποιον τρόπο μπορούν να ενιοποιηθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά και υπάρχουν χώρες στις οποίες ισχύει ένας υψηλότερος ε, πύχης ε, προστασίας των καταναλωτών. παρόλα αυτά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ε, ενιαία αγορά και πρέπει να το έχουμε και αυτό κατά νου. Θέλουμε να καταργήσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν και όχι να δημιουργήσουμε επιπλέον νομικά εμπόδια. Θέλουμε να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες όσον αφορά ε, το εμπόριο στην ενιαία αγορά και ταυτόχρονα θέλουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των πολιτών και των καταναλωτών. Θέλω λοιπόν να σας παροτρύνω να μου υποβάλλετε τα δικά σας σχόλια όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής αυτού του κανονισμού. Αν δεν λάβουμε υπόψη, αν δεν συμπεριληφθούν οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, τα e-books, τα λογισμικά, τα παιχνίδια υπολογιστή και η μουσική, δεν θα έχουμε ε, κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση που θέλαμε. Ε, γιατί θα εξακολουθήσουμε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένο οπτικοακουστικό υλικό στη χώρα μας, χωρίς ωστόσο να έχουμε ταυτόχρονα πρόσβαση στο ίδιο υλικό όταν βρισκόμαστε σε κάποια άλλη ε, χώρα. Η κυρία Ντελβόη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Νομίζω η πρόταση αυτή της Επιτροπής που έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό και άλλου είδους διακριτικές μεταχειρήσεις που δεν δικαιολογούνται και έχουν να κάνουν μόνο με την επικότητα κτλ. Είναι ένα θέμα στο οποίο προσυπογράφω πλήρως, δηλαδή ως προς την όλη προσπάθεια. Σήμερα όμως θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρους των μικρών μικρών επιχειρήσεων και μικρών χωρών. Δύο ζητήματα θέλω να θίξω. Το πρώτο αφορά τις επιχειρήσεις. Ο κανονισμός προβλέπει την υποχρέωση πώλησης σε όλους τους πολίτες που βρίσκονται εντός ένωσης. Ναι, ανάλογα με την μέρημνα που και εσείς εκφράσατε. Πολύ καλά. Αν όμως οι επιχειρήσει πάνε σε άλλη χώρα από αυτήν της κατοικία τους, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να σεβαστούν τους νόμους της χώρα στην οποία πολλούν. Αυτό υποχρεώνει τις μικρές ε, εταιρείε να γνωρίζουν τουλάχιστον 28 διαφορετικές νομοθεσίες. Φαντάζομαι ότι μεγάλες, για τις μεγάλες πολυεθνικές χώρε να πω ονόματα δεν είναι πρόβλημα. Υπάρχει μια υπηρεσία με δικηγόρους, ε, έχουν ε, δυνατότητες να ασχοληθούν με οτιδήποτε προκύψει, αλλά οι μικρές επιχειρήσεις, εφόσον θέλουν να πουλήσουν διασυνοριακά, λένε, αν πρέπει να πληρώσω και για τα δικηγορικά τέλη για 28 διαφορετικές χώρες, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Οπότε πρέπει λίγο να σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να διευκολύνουμε τη ζωή των μικρών επιχειρήσεων αν θέλουμε να ε, ευνοήσουμε το διασυνοριακό εμπόριο. Εδώ μιλάμε για άρση συνόρων αντί να τα καταπολεμούμε. Και δεύτερος προβληματισμός σε ό,τι αφορά τις μικρές χώρες. Και μιλώ εν ε, πλήρη γνώση των πραγμάτων γιατί Έρχομαι από το Λουξεμβούργο και στο Λουξεμβούργο ε, μας αρέσει να αγοράζουμε. Μας αρέσει να αγοράζουμε online και μας αρέσει να αγοράζουμε και από ξένες χώρες, τις γειτονικέ. Ο πολίτης λοιπόν έχει την υποχρέωση να πωλήσει αλλά όχι να παραδώσει το εμπόρευμα. Δεν το, παρα... δεν το βρίσκω φυσιολογικό αυτό. Δηλαδή ζω στο Λουξεμβούργο, παραγγέλνω κάτι στη Γερμανία και πρέπει να επινοήσω μία διεύθυνση κοντά στα σύνορα στη Γερμανία ή στη Γαλλία για να παραλάβω αυτό που παρήγγειλα. Αν το δικαίωμα αγοραπολισίας δεν συνδυάζεται με το δικαίωμα παράδοσης και όλα στο εμπορεύματος της υπηρεσίας, τότε τι νόημα έχει. Ε, με τα σύνορα λοιπόν αυτά πρέπει να πω ότι ειλικρινά ενοχλούμε τα μάλα. Θα ήθελα εδώ να ε, βρεθεί κάποια λύση. Μια λύση γιατί αυτό αφορά ιδιαίτερα στις μικρές χώρες. Και ιδίω τι διασυνοριακές περιοχές, τις παραμεθόριες μάλλον περιοχές των μεγάλων χωρών. Εκεί είναι σημαντικό το τι γίνεται. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κυρία Ντελβό. Ο κύριος Κάντεφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ θα σας τα πω εκ μέρους του κυρίου Γκρόγκε, που είναι ο εισηγητής του ΕΛΚ. Και μιλάμε για το γεωγραφικό αποκλεισμό στην επιτροπή μας. Πρέπει να δούμε τι γίνεται εδώ με τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Για την ε, αγορά που φαίνεται να επιτρέπει, ότι θα, μάλλον θέλουμε να επιτρέπει στους καταναλωτές να αγοράζουν ε, υπηρεσίες και αγαθά σχέτως της εθνικότητάς τους, της υπηκότητάς τους. Εδώ ο γεωγραφικός αποκλεισμός ε, με την διακριτική μεταχείριση προ προς τις τιμές, με τον κατακαιρματισμό της αγοράς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ο κ. Γκρόκε λέει ότι θα πρέπει να είναι σαφές και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές ότι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή. Πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερη νομική βεβαιότητα για το πόσο εφαρμόζονται οι εθνικές νομοθεσίες περί συμβάσεων και ιδίω για τις επιγραμμικές αγοραπολισίες και ότι πρέπει να υπάρχει σαφήνεια για τους καταναλωτές. Στην Επιτροπή μας πρέπει να εργαστούμε για ευθύς λύσεις και τώρα Πρέπει να δούμε τους αποκλεισμού για τον κανονισμό αυτό, ιδίως σε συνδυασμό και με τον τομέα των μεταφορών. Ο κ. Κράγκε ε, ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να συμμετάσχει στη σημερινή συζήτηση, αλλά υπογραμμίζει ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον ε, εισηγητή, τους Σκιώδης και όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους προκειμένου να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση. Ε. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα εισηγήτρια... Ε, και τώρα να δούμε ποιο άλλο θέλει το λόγο, διότι και εγώ θα συμφωνήσω με την συνάδελφο Ντελβό. Γιατί το δικαίωμα παράδοσης πρέπει να συνδυάζεται με το δικαίωμα ε, με την υποχρέωση αγοραπολισίας. Δεν πρέπει να έχουμε εδώ μια κατάσταση και πρέπει να βρεθεί μια λύση αισιόδοξη. Μια λύση που να μπορεί να ικανοποιεί κυρίως τους πολίτες μας. Θέλουμε να διευκολύνουμε τα πράγματα. Στο μέλλον θέλουμε να υπάρχει πρόσβαση Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που παρακολούθησα τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάσατε την έκθεσή σας και στηρίζω αυτή την ιδέα της διεύρυνσης του θέματος και ε, της συμπερίληψης και άλλων υπηρεσιών. Νομίζω ότι για να ξεμπλοκάρουμε την πρόσβαση σε διάφορες επιγραμμικές υπηρεσίες, τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται διαδικτυακά. Και θα μπορούσε αυτό να είναι μια καλή ιδέα. Συνάμα όμως πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο να συνεχίσουμε να σεβόμαστε τα δικαιώματα copyright σε όλη την Ευρώπη, έτσι ώστε οι άνθρωποι που παράγουν προϊόντα και τα οποία διανέμονται στην Ευρώπη να μπορούν να αποκτήσουν χρήματα για αυτά, όπως για παράδειγμα είναι η περίπτωση των καλλιτεχνών. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να εισπράττουν, θα μπορούν να πληρώνονται για τη διανομή αυτών των προϊόντων σε διαδικτυακό επίπεδο. Ζήτησα το λόγο γιατί ήθελα να αναδείξω περισσότερο τα παραδείγματα διακρίσεων για να στηρίξω περισσότερο το επιχείρημά μου γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και να μιλάμε συγκεκριμένα. Τρία είναι τα παραδείγματα με τα οποία δημιουργείται διάκριση λόγω του geo-blocking, γεωγραφικού αποκλεισμού. Έχουμε video content services, υπηρεσίες περιεχομένου βίντεο. Πάρα πολλές εταιρείες παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες στην Ευρώπη. Η Netflix, η HBO είναι μεγάλες επιχειρήσεις συνήθως και αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να είναι διαθέσιμες και να διαθέτουν τα προϊόντα τους, την υπηρεσία τους σε όλα τα κράτη-μέλη, γιατί είναι μεγάλες, έχουν ένα σωρό δικηγόρους που δουλεύουν για αυτές και παρέχουν την υπηρεσία παντού. Τι κάνουν λοιπόν. Εφαρμόζουν μια ταρίφα την ίδια στα διάφορα κράτη-μέλη, ενώ εφαρμόζουν την ίδια το περιεχόμενο στο οποίο επιτρέπουν ε, την πρόσβαση δεν είναι το ίδιο. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, είναι 25 ευρώ το μήνα για περιορισμένο περιεχόμενο, ενώ στη Γαλλία είναι πάλι 25 ευρώ το μήνα με πολύ μεγαλύτερο περιεχόμενο, με πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερο περιεχόμενο. Και αυτό είναι συγκεκριμένο παράδειγμα διάκριση που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή. Άλλο παράδειγμα. Αθλητική σταθμή. Και θα σας δώσω και ονόματα, το Canal Plus Sport, το Eurosport, εδώ. Πληρώνετε για αυτό το περιεχόμενο, πληρώνετε για αυτή την υπηρεσία, μπορείτε να παρακολουθήσετε ορισμένους αγώνες, ορισμένα αθλήματα, αλλά σας απαγορεύεται να παρακολουθήσετε άλλου είδους αγωνίσματα ή αθλήματα ή αγώνες. Για παράδειγμα, ε, διανομή του Champions League. Ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Πληρώνετε για την υπηρεσία, αλλά όταν διανέμετε ειδικό περιεχόμενο δεν έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία. και δεν έχετε δυνατότητα να το παρακολουθήσετε. Ορίστε δύο παραδείγματα διακρίσεων που λαμβάνουν χώρα σήμερα λόγω του γεωγραφικού αποκλεισμού. Και πράγματι, αυτά τα στοιχεία αποκλεισμού επηρεάζουν και τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν, δεν δύνανται να πολεμήσουν τους μεγάλους παίκτες, γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση επαρκή για να ε, ε, ανοίξουν οι αγορές, να έχουν πρόσβαση σε όλα τα κράτη ένα προς ένα, ενώ οι μεγάλες εταιρείες είναι παρούσες παντού και μπορούν να ανοίξουν την πρόσβαση σε όλες τις αγορές. Ε, μία δεύτερη αρνητική επίπτωση του γεωγραφικού αποκλεισμού είναι η εξή. Λυσμονούμε πολύ συχνά ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες που μετακινούνται από τη μία ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη θα πρέπει να κρατήσουν και χρειάζονται να κρατήσουν βασικά, ήδη το χρειάζονται, ε, πιο στενή πρόσβαση με τα τεκτενόμενα στη δική τους χώρα προέλευσης και ε, δυσκολεύονται να έχουν στενή επαφή, δυσκολεύονται να ε, ε, έχουν πρόσβαση στι ίδιε και τηλεοπτικέ, για παράδειγμα, υπηρεσία με του συμπατριώτε του. Δεν βλέπουν την ίδια τηλεόραση, δεν μπορούν να δουν τα ίδια κανάλια που βλέπαν στην πατρίδα του. Και λέγεται ότι στηρίζουν τη χώρα προέλευσης και το καθεξής. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε και αυτούς που ζουν σε άλλες χώρες στην Ευρώπη και θέλουν να διατηρήσουν την επαφή με την πατρίδα τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεμπρετού θα ήθελε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σε αυτό το όμορφο πλαίσιο που μας παρουσιάζεται από τη στιγμή που αντιλαμβάνομαι ότι όλοι είναι υπέρ της κατάρρισης του γεωγραφικού αποκλεισμού ε, εξ ονόματος της δημιουργίας μιας μεγάλης και πανέμορφης ψηφιακής αγοράς, εγώ θα είμαι η κοιλίδα που θα στοιχιώσει κάπως το τοπίο, διότι επιθυμώ ότι πρέπει να επιθυμώ να παραμείνει ο γεωγραφικός αποκλεισμός για να διατηρηθούν οι ιδιαιτερότητες της εθνικής υπηρεσίας ε, παροχής περιεχομένου. Αυτό το οποίο με ενοχλεί είναι ότι συνήθως επικαλείστε τα επιχειρήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες υποτίθεται ότι δεν έχουν τα μέσα να έχουν πρόσβαση στην πραγματικότητα των 28 ε, κρατών μελών. Στην πραγματικότητα όμω, εσεί εξυπηρετείτε το παιχνίδι των μεγάλων επιχειρήσεων, γιατί μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες θα επωφεληθούν καταρχάς από την κατάρριξη του γεωγραφικού αποκλεισμού και τα τεράστια λόμπι τους θα διωγγωθούν ακόμα περισσότερο δεν είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις των οποίων το όνομα αναφέρεται, είναι οι μεγάλες. Netflix δεν είναι. Η Netflix και το Eurosport δεν είναι καμία μικρομεσαία επιχείρηση που κινδυνεύει. Ακούγοντάς σας δεν είμαι καθόλου πεπισμένος για το ότι είναι σκόπιμο να καταργηθεί ο γεωγραφικός αποκλεισμός εξ και για χάρη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καθόλου δεν με πείθεται. Ελπίζω να μπορέσουμε να σας πείσουμε στο μέλλον, λέει η Πρόεδρος. Και θα βρούμε ορθά παραδείγματα με μικρές επιχειρήσεις. Η συζήτηση μόλις τώρα ξεκίνησε. Θα πάμε και πιο πέρα. Ε, μιλώντας γαλλικά, κυρία μου, ήδη διανύσατε τη μισή διαδρομή μέχρι να με πείσετε τελείως. Και θα συνεχίσω, κύριε Λεμπρετού. Θα ζητήσω από τον συνάδελφο να προεδρεύσει, γιατί πρέπει να φύγω. Είναι ο κύριος Φως. Um, λοιπόν, θα προχωρήσουμε και θα περάσουμε στο σημείο 31. Μιλάμε για την εφαρμογή της οδηγίας 2004 34 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την παραπληκτική ευθύνη και την πρόληψη ε, και την αποζημίωση σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας, τη γνωστή οδηγία ELD. Έχουμε λοιπόν μια ανταλλαγή απόψεων με την Κομισιόν. Θα ήθελα καταρχάς να ε, καλέσω τους εκπροσώπους της Κομισιόν να κάνουν μια σύντομη παρουσίαση της έκθεσης του Απριλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Ο κύριος Hans Λοπάτα έχει προσκληθεί. Πού είναι? Εκεί. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Έχετε το λόγο Παρακαλώ σας ακούμε. Thank you. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ευρωβουλευτές. Είμαι εδώ μαζί με τον συνάδελφό μου κύριο Χάνς Λοπάτα για να σας παρουσιάσουμε την έκθεση της ε, Κομισιόν και την αξιολόγηση REFIT της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη καθώς και να σας παρουσιάσω τις ε, δραστηριότητες που έχουν ε, προγραμματιστεί για το περίοδο 2017-2020. Να ξεκινήσω με την έκθεση. Evaluation. Η αξιολόγηση της οδηγίας για την προβληματική ευθύνη ε, ακολούθησε δύο διαδικασίες. Πρώτον ήταν η, το άρθρο 18 το της ίδιας της οδηγίας, το οποίο προβλέπει ότι η Κομισιόν θα κάνει έναν απολογισμό σε σχέση με την εφαρμογή της ε, εν λόγω οδηγίας. Η δεύτερη διαδικασία ήταν το πρόγραμμα REFIT της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του οποίου η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να αξιολογήσει την καταλληλότητα για το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε της νομοθεσίας ε, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνεκτικότητα και την πρόσθετη αξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί λοιπόν ήταν οι λόγοι για τους οποίους διοργανώθηκε αυτή η αξιολόγηση REFIT. Οι κύριες πηγές ήταν οι εκθέσεις ε, τις οποίες παρήχαν τα κράτη-μέλη σχετικά με την εφαρμογή της ε, ELD και αυτές οι εκθέσεις ε, ξεκίνησαν το 2013 και εμείς με δική μας πρωτοβουλία εκπονήσαμε μια σειρά από μελέτες τα έτη 2013-2014 όπως είχε προβλεφθεί εξ αρχής. Επίσης η Κομισιόν έλαβε υπόψη της τα συμπεράσματα της προηγούμενης έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη που είχε διεξαχθεί το 2010 καθώς και τα σχόλια που ε, λάβαμε μέσω των συναντήσεών μας με κυβερνητικούς αξιωματούχους στο πλαίσιο της Επιτροπής ELD αλλά και με ευρύτερα τους εμπλεκόμενους φορείς που ε, θίγονται από την ELD. Το βασικό ερώτημα λοιπόν ήταν αν η Οδηγία 37 για την οικονομική, ε, ε, για την περιβαλλοντική ευθύνη είναι κατάλληλη σε σχέση με, την, ε, με τον στόχο για τον οποίο είχε ψηφιστεί και αν έχει επιτύχει τους σκοπούς για τους οποίους είχε θεσπιστεί. Να περάσω τώρα στα βασικά πορίσματα και εδώ το καλύτερο θα ήταν να σας παραθέσω τα λόγια της ίδιας της έκθεσης που αναφέρει ότι τα συνολικά πορίσματα από τις πληροφορίες και τα δεδομένα επιβεβαίωσαν το συμπέρασμα της προηγούμενης έκθεσης του Οκτωβρίου 2010 για μια ε, σημαντική ποικιλομορφία μεταξύ των ε, διαφόρων κρατών μελών. Παρά τις προσπάθειες που είχαν αναλυφθεί έως εκείνο το στιγμή από την Κομισιόν και τις ομάδες των ε, εμπλεκόμενων φορέων να δημιουργηθεί ένας, ε, ένα πλαίσιο ίσων όρων ε, μέσω μη νομοθετικών μέτρων, όχι μόνο η μεταφορά στο εθνικό δίκτυο, αλλά και η εφαρμογή αυτής της οδηγίας ε, ποικίλει σημαντικά από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Και γι' αυτό το λόγο αυτή, αυτός ο κατακαιρματισμός όσον αφορά την περιβαλλοντική ευθύνη συζητήθηκε ε, σε πολλές, ε, και εξετάστηκε σε πολλές από τις ε, μελέτες που αφορούσαν την αξιολόγηση της ELD. Όπως βλέπετε το βασικό πόρισμα ήταν πραγματικά αυτό το μοσαϊκό όσον αφορά την εφαρμογή. Ποιοι ήταν οι κύριοι παράγοντες που προσδιορίστηκαν στην έκθεση REFIT για την ELD. Πρώτος παράγοντας ήταν η συνεχιζόμενη χρήση προϋπάρχουσας εθνικής νομοθεσίας σε σχέση με την περιβαλλοντική ευθύνη αντί της οδηγίας ELD ή ε, σε συνδυασμό με αυτήν. Επίσης, υπήρξε σημαντικό, ε, ε, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε ένα πολύ μεγάλο, πολύ ψηλό όριο σημαντικότητας όσον αφορά την, τις, τις περιβαλλοντικές ζημίες. Επίσης, υπάρχουν διαφορετικές ε, διαφορετικό επίπεδο ενδιαφέροντος των εμπλεκόμενων φορέων όσον αφορά την συνεργασία τους με τις ε, αρμόδιες αρχές. Διαπιστώσαμε ότι υπήρξαν ε, διαφορές όσον αφορά τις υποχρεώσεις των αρμοδίων αρχών να παρέχουν μέτρα αποζημίωσης και Επίσης υπήρξε μεγάλη ετερογένεια όσον αφορά την ευαισθητοποίηση γύρω από την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη, όσον αφορά τις, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει από τους φορείς εφαρμογής αλλά και από το, ε, από το κοινό. Όλοι αυτοί οι παράγοντες λοιπόν συνέβαλαν σε αυτήν την πολύ μεγάλη ποικιλομορφία ανάλογος της κατάστασης που επικρατεί σε κάθε κράτος μέλος. Ποια ήταν η ανταπόκριση της Κομισιόν σε αυτά τα πορίσματα. Ήταν ε, προφανώς τα, οι δράσεις που θα αναλυθούν τα επόμενα χρόνια, η προοπτική που δίνεται. Πρώτον, ε, έχουμε ξεκινήσει ένα πολυετές σχέδιο εργασίας για την ELD για την περίοδο 2017-2020 που βασίζεται στα συμπεράσματα και στις συστάσεις της έκθεσης ELD και της αξιολόγησης REFIT Οπότε θα υπάρξει ένα πολιετές σχέδιο δράσης ε, που θα καταρτιστεί σε συνεργασία από κοινού μεταξύ ε, από τα κράτη-μέλη και από την Κομισιόν. Αυτό το σχέδιο δράσης πρόκειται να ε, εγκριθεί στην επόμενη συνάντηση των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών τον Φεβρουάριο του 2017 και προφανώς θα υπάρξει η θα υπάρξει και εξωτερική τεχνική βοήθεια όσον αφορά την εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράσης του πολιετούς. Ποιοι θα είναι οι κύριοι τομείς εργασίας, οι προτεραιότητες δηλαδή σε αυτό το πολιετές ε, πρόγραμμα ε, δράσεων τα επόμενα χρόνια. Πρώτον, υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί η βάση των ενδείξεων σχετικά με την ε, αξιολόγηση της ELD, δηλαδή θα υπάρξει ένα καλύτερο πλαίσιο για την αξιολόγηση, το οποίο θα αναπτυχθεί του χρόνου, στη συνέχεια θα δοκιμαστεί και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2018, ένα πλαίσιο αξιολόγησης λοιπόν. Επίσης θέλουμε να ε, επικεντρωθούμε στην περαιτέρω ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων και μέτρων για να υπάρξει μια ολοένα και πιο ομοιογενής εφαρμογή της οδηγίας και αυτό πράγματι αφορά τόσο την ανάπτυξη μιας κοινή αντίληψης των βασικών ενιών και όρων, να υπάρξει δηλαδή μια σταθεροποίηση γύρω από αυτό το θέμα μέσω της ε, περαιτέρω επεξεργασίας και της εφαρμογής μιας ε, έννοιας ε, δημιουργίας ικανοτήτων ολοκληρωμένης. Για παράδειγμα, στο παρελθόν έχουμε παράσχει μια εκπαιδευτική μονάδα στα κράτη-μέλη σχετικά με την EOLD, την οποία και θα επεκτείνουμε στο μέλλον. Άλλο σημείο που μας ενδιαφέρει είναι ε, η εξασφάλιση ε, επαρκών, επαρκούς και ζήτησης για την οικονομική ασφάλεια προκειμένου να καλύπτονται οι ευθύνες που προκύπτουν από την ELD. Φυσικά ε, εδώ σημαντικό είναι και η δημοσιονομική ασφάλεια που, παρέχεται ε, γιατί αν, υπάρχει, αν προβλέπεται ευθύνη αλλά δεν υπάρχει τρόπος χρηματοδότησης της, προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει να ελέγξουμε δηλαδή και να μετρήσουμε την ζήτηση και την οικονομική ασφάλεια σε όλα τα κράτη-μέλη. Καθώς λοιπόν πρόκειται για ένα σχέδιο δράσης της Κομισιόν και, και των κρατών μελών, προφανώς ε, παρέχουμε και ορισμένες συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Να σας δώσω λοιπόν μια ε, συνοπτική παρουσίαση ποιες θα είναι αυτές οι συστάσεις. Πρώτον θέλουμε τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες εφαρμογής με δραστήριες πρωτοβουλίες και εδώ έχουμε μια σειρά από καλά παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές όπως είναι τα καθοδηγητικά έγγραφα, η εκπαιδευτική κύκλη, τα ηλεκτρονικά εργαλεία για την ανάλυση κινδύνου, ε, έχουμε μοντέλα για την οικονομική ασφάλεια. Υπάρχουν μια σειρά από μέτρα και προσπάθειες λοιπόν σε διάφορα κράτη-μέλη, φυσικά με πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Επίσης θέλουμε να ενισχύσουμε την ανταλλαγή ε, εμπειριών, διοικητικών και βέλτιστων πρακτικών και να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη όσον αφορά τη δημιουργία ικανοτήτων. Επίσης, θέλουμε σε πνεύμα συνεργασίας να εξετάσουμε την ερμηνεία βασικών διατάξεων της οδηγίας και συγκεκριμένα όσον αφορά ε, το θέμα της, ε, της σημασίας, της σημαντικότητας, αυτό το όριο σημαντικότητας το οποίο έχει ερμηνευτεί με αρκετά ευρύ θα έλεγα τρόπο. Είναι λοιπόν μία από τις προτεραιότητες μας να ενιοποιήσουμε κατά κάποιον τρόπο την ερμηνεία που δίνεται σε τέτοιους όρους. Επίσης, Για την καλύτερη εφαρμογή της ELD χρειαζόμαστε καλύτερα στοιχεία, περισσότερες γνώσεις και για αυτό το σκοπό φυσικά χρειαζόμαστε τη συνεργασία των κρατών μελών αλλά και των δικών μας υπηρεσιών προκειμένου να καταγράφονται και να καταχωρίζονται τα περιστατικά και οι υποθέσεις που υπάγονται στην ELD ε, σε επίπεδο εθνικής αλλά και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τα αντίστοιχα μητρώα. Όχι μόνο για τη βάση ε, των, γνώσεων, αλλά και για λόγους διαφάνειας. Και να συνεχίσουμε φυσικά την συλλογή δεδομένων ανακράτος μέλος σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας, ιδίως ε, στα κράτη-μέλη ε, που, ε, από τα οποία μπορούμε να αντιλήσουμε θετικά παραδείγματα και διδάγματα σχετικά με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Αυτά ως επισκόπηση νομίζω ότι τήρησα και τον χρόνο που μου δώσατε και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επισκόπηση και τώρα προσκαλώ τον εισηγητή μας, την εισηγητριά μας για την έκθεση σε σχέση με την υλοποίηση, την κυρία Φεράρα να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή για αυτή την πρώτη παρουσίαση της έκθεσης. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτήν την ε, έκθεση. Ε, και για τις διαδικασίες επαλήθευσης και αξιολόγησης με μια σειρά μελετών που έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την ευχαριστούμε. Η τελευταία μόλις μας παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Γιούρη. Από όσα λέγονται λοιπόν σε αυτά όλα τα κείμενα, η κατάσταση είναι σχετικά ε, μη ικανοποιητική, όχι μόνο ως προς την ε, ίδια την υλοποίηση, αλλά και τα εργαλεία που προβλέπει η οδηγία και την αποτελεσματικότητά τους ε, για να επιτευχθούν επιδιωκόμενοι στόχοι. Είδαμε ότι υπάρχει μια διαδικασία υλοποίησης αργή, ετερογενής, και δεν υπάρχει συμμόρφωση από πολλές ε, απόψεις ε, όσα προβλέπονται από την Επιτροπή. Και η οδηγία πλαίσιο στο νομοθετικό επίπεδο δεν ε, έχει προβλέψει κατά τις 100% ομοιογένεια και ομοιομορφία στην υλοποίηση. Πολύ λίγα κράτη, μόνο δύο, η Ουγγαρία και η Πολωνία, το 86% όλων των υποθέσεων, των ζημιών που έχουν ε, επισημανθεί, ε, ε, έχουν καταφέρει να υλοποιήσουν σωστά. Άρα πρέπει να καταλάβουμε και τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν αυτές οι ανισότητες, αυτές οι διαφορές μεταξύ των περιπτώσεων. Φταίει η εθνική νομοθεσία, φταίει ο αριθμός των ελέγχων που γίνονται, που δημιουργούνται, ε, είναι μια ιδιαιτερότητα ε, που είναι ενδογενή στην ε, περίπτωση του συγκεκριμένη χώρα, τη περιοχή. Επίση, κάτι άλλο που μα ε, επεσήμανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το τι γίνεται με την περιβαλλοντική σκοπιμότητα και ένα κράτο μέλο. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να συνάδει και με την εθνική νομοθεσία και με τις διεθνείς συμφωνίες, αλλά αυτό δεν γίνεται πάντοτε με απόλυτη συνοχή και συνεκτικότητα. Εκεί ε, προσκρούει η ομαλή υλοποίηση της οδηγίας. Εν γέννη, τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με τις παρεμβαλλοντικές συνθήκες των κρατών μελών είναι κατακαιρματισμένα, είναι αποσπασματικά. Εδώ λοιπόν για να αξιολογήσουμε σωστά την αποτελεσματικότητα της οδηγίας και να είναι και αξιόπιστα τα στοιχεία που διαθέτουμε πρέπει και από επιστημονικής και νομικής πλευράς να έχουμε καλύτερα στοιχεία. Τους επόμενους μήνες μαζί με τους με τον συνάδελφο Γιάβορα από την Επιτροπή ΕΝΒΗ, θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά για την έκβαση αυτή. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να παροτρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην όλη προσπάθεια αναθεώρηση τη οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη. Ε, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σε ποιε πτυχέ τη οδηγία θα πρέπει να αναλάβουμε δράση λόγου χάρη για το πεδίο τη περιβαλλοντική ευθύνη, εκεί να καλύψουμε τα διάφορα κενά, την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών αρχών, προκειμένου να προβλέψουμε και να προλάβουμε τι διάφορε ζημιέ, στην ίδρυση, στην δημιουργία εθνικού μητρώου ε, σε εθνικό επίπεδο για του ε, φορεί που δραστηριοποιούνται σε κάθε χώρα, προκειμένου να διευκολύνουμε και την δουλειά των ελεγκτικών αρχών και να υπάρχει και μια διαδικασία πρόληψης. Επίσης η υποχρεωτική καταγραφή και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό η προστασία του περιβάλλοντος από ζημιές που προκύπτουν από μηχανική δραστηριότητα. Και εδώ ε, η Επιτροπή θα πρέπει να κοιτάξει μια βελτίωση στην ε, εκτέλεση των πόρων, ώστε να βελτιωθεί και η συνολικά υλοποίηση της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη. Υπάρχουν ε, κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες και πρέπει να λαμβάνονται σοβαρότατα υπόψη. Πάντως, είναι μια χρήσιμη ευκαιρία, όπως έλεγα, για να ξαναορίσουμε και την όλη έννοια της παραπλανητικής ζημίας. Δηλαδή να δούμε ποια είναι τα όρια ανά των οποίων καθορίζεται αυτή η πραγματική ζημία. Και επίση ένα κατάλογο εξαιρέσεων. Ένα κατάλογο εξαιρέσεων που προβλέπει η οδηγία που ίσω πρέπει να αναθεωρηθεί και αυτό. Έπειτα υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα ήθελα να ζητήσω. Είναι ευκαιρία που είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λύσουμε κάποιε απορίε. Στην δεύτερη έκθεση υλοποίηση για την περιβαλλοντική ευθύνη, τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Ιταλία από το 2013 έχει εντοπίσει μόνο 17 περιπτώσει παραβίαση τη οδηγία. Ταυτόχρονα όμω λέει ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλε χίλιε ε, περιπτώσει για τι οποίε θα ήταν υπεύθυνη η Ιταλία για κάποια ζημιά. Ε, θα μπορούσατε να το διευκρινίσετε λιγάκι αυτό. Σε τι αναφέρεστε, Τι είναι οι Ιταλέ χίλιε είναι τίποτα σε εκδίκαση, είναι πρόβλεψη έτσι χονδρική, τι είναι. Έπειτα, κατά την άποψη της Επιτροπής, θα μπορούσε να επεκταθεί το πεδίο της οδηγίας, καλύπτοντας ένα γενικότερο πλαίσιο, εντός του οποίου εντάσσεται και άλλες πτυχές, όπως η ρήπανση των ε, υδάτων από καύσιμα, από όσα προβλέπουν οι διεθνεί μα συμφωνίες και σε συνδυασμό με την εθνική νομοθεσία και σε συνδυασμό με, την, ε, διεθνή, με τους διεθνείς κανόνες. Ανάλογα από ποια άποψη εκλαμβάνεται η οδηγία. Και ως προς την τωρινή κατάσταση και τα αποσπασματικά στοιχεία που έχω μεταξύ των κρατών μελών, Χρειάζεται ένα σύστημα ελέγχου, ένα σύστημα ελέγχου για τα περιβαλλοντικά, για να δούμε αν είχε θετικέ επιπτώσεις η οδηγία. Μα ενδιαφέρει λοιπόν να δούμε αν έχουμε μελέτες, δεδομένα για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στις καλές πρακτικές, αυτές τις οποίες αναφέρονται για ορισμένα κράτη-μέλη. Εν τέλει, στην έκθεση τη 14η Απριλίου 2016, κατά την ελοπίση τη οδηγία λέγεται, εντοπίστηκαν περιπτώσει μη συμβατότητα, μη συμμόρφωση. Και όλα αυτά ε, συνεχίζονται ω σήμερα. Από πού προκύπτουν όλα αυτά, Υπάρχουν λόγοι οι οποίοι διαρκώ επαναλαμβάνονται, υπάρχουν συγκεκριμένε αμέλειε ή πλημελεί ε, ε κινήσει από την πλευρά των κρατών μελών. Εκεί θέλουμε διευκρίνηση. Πρέπει να το καταλάβουμε καλύτερα. Νομίζω η δουλειά μας θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Θα εμπλακούμε αναγκαστικά πάρα πολύ, θα πρέπει να ανασκουμποθούμε για να έχουμε επικοδομητικά αποτελέσματα, αποτελέσματα τα οποία ε, λόγω και του χαρακτήρα του θέματος να μπορέσουν να φέρουν κάποια θετικά αποτελέσματα. Και βάσει της νομοθεσίας, βάσει της έκθεσης υλοποίησης, ίσως να χρειαστεί και μία ε, αποστολή, να χρειαστούν και κάποιες επισκέψεις για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων στοιχείων. Με την υποστήριξη όλων αυτών των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας, λοιπόν, νομίζω θα μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρα στην σύνταξη αυτής της έκθεσης με τρόπο καλό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Λάουρα Φεράρα για την έκθεση και την επισκόπηση. Και πριν προχωρήσουμε, να ζητήσω από τους σκιώδεις εισηγητές να μου πούν εάν θέλουν το λόγο και αν θέλουν να σχολιάσουν για το θέμα αυτό. Δεν βλέπω κανέναν. Οπότε, Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό ο κύριος Γιάγορα από την Επιτροπή περιβάλλοντο Σύνησε στην επόμενη τη έκθεση αυτή. Θα ήθελα και εσεί να μα κάνετε μια σύντομη δήλωση για το όλο θέμα. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες ιδέες για την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας από την περιβαλλοντική σκοπιά, από τη σκοπιά της Επιτροπής για το περιβάλλον. Είναι σαφές από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι αρκετά τα προβλήματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και τη θέση σε ισχύ και της, της Πολλέ διαφορές υπάρχουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση τη οδηγία στο εθνικό δίκαιο, αλλά και στη συνέχεια σε ό,τι αφορά ε, την εφαρμογή αυτής και ω εκ τούτου δεν είναι παιχνίδι επίση ώρε, δεν είναι ίδιες οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομικοί παράγοντε, οι επιχειρήσει, οι εταιρείε. Και αυτό σαφέστατα είναι κατά της ε, ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Και συμφωνώ απολύτως με τα συμπεράσματα της ε, Επιτροπής. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικά μέτρα για να βελτιώσουμε τη θέση σε ισχύ και την εφαρμογή της οδηγίας. Ορισμένες ε, Ορισμένα προβλήματα ήδη προκύπτουν από την οδηγία. Μπορεί να βελτιωθεί η οδηγία αυτή και θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερις τομείς όπου κατά τη γνώμη μου θα χρειαζόντουσαν ε, βελτιώσεις. Θα πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, να επαναπροσδιορίσουμε την περιβαλλοντική ζημία και να διευκρινίσουμε το κατόφλι σημασίας ή σημαντικότητας, να καταργήσουμε τις παρεκκλήσεις που μας οδηγούν τελικά στη δημιουργία ενός μοσαϊκού συστημάτων και μοσαϊκού παραβάσεων. Αυτά καταρχάς. Δεύτερον, θα πρέπει οι φορείς εκμετάλλευσης να είναι υπόλογοι για οποιαδήποτε περιβαλλοντική ζημία ή βλάβη, ακόμα και για τη ζημία στη βιοποικιλότητα. Ε, πρέπει να υπάρξει σύμπνοια με το παράρτημα 3. Ε, πολλές φορές ε, αξιοποιούνται τέτοιου είδους διατυπώσεις στην οδηγία για να διαλάθουν τις περιβαλλοντικές τους ευθύνης. Τρίτον, θα πρέπει να έχουμε δυνατότητα επιθεώρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε κρατικό επίπεδο, να ενισχυθούν τα κρατικά συστήματα επιθεώρησης και σώματα επιθεώρησης, αλλά υπάρξει και ευρωπαϊκό για να έχουμε τακτική παρακολούθηση των βιομηχανικών τοποθεσιών και με, τόπων, εγκαταστάσεων. Και τέταρτον, θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλο χρηματοδοτικό όργανο να διαμορφωθεί, υποχρεωτική περιβαλλοντική ασφάλιση, με εναρμοντισμένο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη, υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις, για όλα τα κράτη-μέλη, σε ένα παιχνίδι επίησης όρης, για να έχουν οικονομική ευθύνη. Και Από τη στιγμή που υπάρχει ένα εργαλείο για το μοίρασμα των κινδύνων ε, για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο απευθύνεται στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω φυσικών καταστροφών, θα πρότεινα να υπάρξει αντίστοιχο εργαλείο διευκόλυνσης ε, για βιομηχανικές καταστροφές, το οποίο να πληρώνει η βιομηχανία, για να διασφαλίσουμε ότι ο, θα στηριχθεί αρχή σύμφωνα με την οποία ο πληρώνει, ότι θα εφαρμοστεί και στην πράξη. Κάθε φορά που προκύπτει βλάβη και πλήγμα στο περιβάλλον. Να έχουμε ένα σύστημα σε πολλαπλά επίπεδα, υποχρεωτικά ε, ασφαλιστικά καθεστώτα ε, ασφάλιση για περιβαλλοντικές καταστροφές συγκεκριμένη διευκόλυνση για δημιουργία Ταμείου Αντιμετώπισης Βιομηχανικών Καταστροφών και ενίσχυση της επιθεώρησης των εγκαταστάσεων των βιομηχανικών. Όλα αυτά μας βοηθούν ε, να εφαρμόσουμε την αρχή «Ορυπαίνων πληρώνει». Ε, σε αυτού του τομεί θα μπορούσαν να επέρθουν βελτιώσει στην οδηγία και εμεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντο θα πράξουμε τα δέοντα, θα πράξουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, ό,τι καλύτερο για να ασκήσουμε πηγή και ο κανονισμός ευρωπαϊκός να πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, όπου επιτέλους θα πληρώνουν αυτοί που προκάλεσαν τις περιβαλλοντικές ζημίες και όχι το κράτος ή ο φορολογούμενος. Ευχαριστώ πολύ. σε ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ να ζητήσω συγγνώμη από τους προσκεκλημένους μας, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Δώστε μας λίγο χρόνο ακόμα να ακούσουμε τον συνάδελφο, ένα τελευταίο μιλητή και να ζητήσω συγγνώμη και από τον κύριο Χρυσόκονο για την καθυστέρηση της έναρξης του εργαστηρίου του. Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε εν συντομία γρήγορα τα προηγούμενα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Ίσως η Επιτροπή με τον εισηγητή να μπορέσουν να διευκρινίσουν το ζήτημα διμερός, γραπτός, όπως προτιμάτε η ΜΕΝ και η ΔΕ, για να μην καθυστερήσουμε περισσότερο. Έτσι δεν είναι. Και εσείς έχετε ήδη απευθύνει ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκτός μικροφώνου η ομιλήτρια. Είναι αυτό εφικτό? Ναι, συγγνώμη. Εάν δεν υπάρχει χρόνος τώρα βεβαίως και μπορούμε να έχουμε διδημερή ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της γραπτής διαδικασίας με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Καλώς. Ευχαριστώ όλους. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο τελευταίος ομιλητής για το θέμα αυτό, ο κύριος Λεμπρέτου. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα είμαι σύντομος γιατί ο χρόνος πιέζει. Αυτή η οδηγία είναι ένα σημαντικό κείμενο γιατί ε, έχει σκοπό να εξασφαλίσει την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον και να τα, τις προλάβει. Συμφωνώ με την αρχή ότι ο Ριπένον πληρώνει, είναι αυστηρή αρχή αλλά ε, ε, επιβάλλεται και θα πρέπει να δούμε πώς εφαρμόζεται η οδηγία αυτή. Και εδώ διαπιστώνω και υποχρεούμε να το πω ότι ο απολογισμός της εφαρμογής της οδηγίας είναι απογοητευτικός. Πάρα πολλά κράτη έχουν ε, ε, κρατήσει αρχαία νομοθεσία, πεπαλαιωμένη και απαξιωμένη. Άλλοι έχουν περιβαλλον τικές προβλέψεις εξαιρετικά αυστηρές, διαπιστώνω ότι το σημείο κίνησης ήταν ερωτηματικό εξ αρχής, γιατί τέσσερα κράτη είχαν ενσωματώσει την οδηγία τηρώντας την αρχική προθεσμία, άλλα κράτη είχαν προβάλει ισχυρές αντιστάσεις. Σε κάθε περίπτωση οι δύο εισηγητές έκαναν εξαιρετική δουλειά και θα ήθελα να του συγχαρώ. Σπάνια έχω ακούσει τόσες πολλές προτάσεις και ε, στην, όσο άκουσα στην έκθεση της κυρίας Φεράρα και στην έκθεση του συναδέλφου από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Έχω ένα ερώτημα και ελπίζω να μου απαντήσετε γραπτό, που έχει να κάνει με διάφορες χώρες συμπεριλαμβανομένε τη Γαλλία. Σε μία από τι εκθέσει διάβασα ότι ορισμένες χώρες και η Γαλλία απέκλεισαν από το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία του αεροψεκασμού σε ό,τι αφορά την διαχείριση των αποβλήτων. Είναι κάτι το σοβαρό αυτό. Δεν είναι, δυσκολεύομαι να το εκτιμήσω. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε η δική σας ανάλυση τι πιστεύει. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την τελευταία παρέμβαση και με αυτά ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα. Εύχομαι καλή επιτυχία στο εργαστήριο που θα διοργανωθεί αμέσως μετά Ξαναζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό σας βράδυ. Αγαπητοί συμμετέχοντε. με μεγάλη μου χαρά σα ε, καλωσορίζω εδώ, σε αυτό το εργαστήριο για την εφαρμογή του, της οδηγίας για τη δημοσιολάβηση που ε, οργάνωσε το Τμήμα Πολιτικής έπειτα από ε, ε ε, μας. Μπορεί να χρησιμεύσει η διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ε, μέσω προσαρμοσμένης ε, προσαρμοσμένων υπηρεσιών στα συμβαλόμενα ή αντιμαχόμενα μέρη. Πριν από την υιοθέτηση της οδηγίας υπήρχαν μορφές διαμεσολάβησης όπως ε, ε, η ε, Οδηγία 2013 κάθετος 11 για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και ο κανονισμός 524 κάθετος 2013 για, τις, για την επίλυση διαφορών, επιγραμμικών διαφορών. Θα ήθελα επίσης να, να ευχαριστήσω για την παρουσία τους τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Συμβολογράφων της ε, ε, Ευρώπης που έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους για το έργο μας. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Georg Χάιμπα από την Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να μας παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία της έκθεσης της Κομισιόν για την εφαρμογή ε, της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση. Έχετε 15 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ευχαριστώ, να ευχαριστήσω πολύ που προσκαλέσατε την Κομισιόν για να σας παρουσιάσω αυτή την έκθεση. Θα επικεντρωθώ στα βασικά σημεία, καθώς ε, φαντάζομαι ότι πολλοί από εσά έχετε ήδη διαβάσει την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Ποιες ήταν οι πηγές πληροφόρησής μας. Ε, τρεις θα ήθελα να αναφέρω. Εκπονήσαμε μια μελέτη σχετικά με την εφαρμογή της ε, οδηγίας το 2013 και την ε, επικαιροποιήσαμε το 2016. Κάναμε μια μονοήμερη συζήτηση ε, στο πλαίσιο του δικτύου δικαιοσύνης για αστικά και εμπορικά ε, ζητήματα, όπου συζητήσαμε τα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας στα κράτη-μέλη και επίσης Υπήρξε μια διαβούλευση πέρσι όπου ζητήθηκε από τους εμπλεκόμενους φορείς να υποβάλουν τα σχόλιά τους σχετικά με την εκτέλεση και την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Η έκθεση της Κομισιόν γενικά συμπεραίνει ότι συνολικά η οδηγία έχει ε, προσφέρει προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση των εθνικών νομοθετών όσον αφορά την αξία ε, της, διαμεσολε... διαμεσολάβησης και η οδηγία επίσης είχε πολύ θετικά αποτελέσματα σε κράτη-μέλη που όμως ε, το, ο βαθμός που επηρέασε η οδηγία ε, σχετίζεται με το σύστημα το προϋπάρχων Σε 15 κράτη-μέλη προϋπήρχε ήδη διαμεσολάβηση. Εκεί οι αλλαγές που επέφερε η οδηγία ε, ήταν κάπως πιο περιορισμένη. Σε εννιά ε, χώρες υπήρχαν κατακαιρματισμένοι κανόνες από εδώ και από εκεί ή ε, επαφιόταν στους, σε ιδιωτικούς φορείς. Σε αυτές τις χώρες, ωστόσο, η οδηγία επέφερε μεγάλες αλλαγές. Σε τέσσερα κράτη-μέλη, για πρώτη φορά ε, υπήρξε διαμεσολάβηση με βάση ε, αυτή την οδηγία και φυσικά εκεί είναι, είναι τα κράτη-μέλη στα οποία η οδηγία επέφερε τις σημαντικότερες αλλαγές. Επίσης, ε, συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες όσον αφορά τα εθνικά συστήματα διαμεσολάβησης στην πράξη. Αυτές οι δυσκολίες σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη μιας κουλτούρας διαμεσολάβησης, της έλλειψης γνώσεων για το πώς θα πρέπει να γίνεται ο χειρισμός των διασυνοριακών υποθέσεων, η χαμηλή ευαισθητοποίηση και ε, ο, ο ανεπαρχής τρόπος λειτουργίας των μηχανισμών εξασφάλισης της διαμεσολάβησης. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι λοιπόν. Ε, ε, για την καλή ή τη λιγότερο καλή εφαρμογή διαφόρων άρθρων και εδαφείων της οδηγίας. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στα σημαντικότερα που θα τεθούν και στο επίκεντρο του σημερινού μας εργαστηρίου. Πρώτον είναι το πεδίο ισχύω της οδηγίας και το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει την οδηγία και για εσωτερικές υποθέσεις, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Μόνο τρία κράτη-μέλη ε, περιόρισαν την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο μόνο στις διασυνοριακές υποθέσεις. Πρόκειται προφανώς για ένα αποτέλεσμα το οποίο εμείς το, το, το χαιρετίζουμε βεβαίως, γιατί έτσι ο αριθμός των υποθέσεων που επιλύονται μέσω διαμεσολάβηση ε, είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι αν περιοριζόταν μόνο στι διασυνοριακέ υποθέσει. Η δεύτερη πτυχή που θέλω να αναφέρω είναι το ζήτημα της ποιότητας, των προδιαγράφων ποιότητας ε, για τη διαμεσολάβηση. Ε, εδώ, ιδίως στην δημόσια διαβούλευση, αναδείχθηκαν ε, κάποια επιχειρήματα υπέρ και κάποια επιχειρήματα κατά της εκπόνησης ευρωπαϊκών προδιαγραφών ποιότητας. Είναι ένα ζήτημα αμφιλεγόμενο δηλαδή με άλλα λόγια. Ωστόσο, οι απαντήσεις που λάβαμε στο πλαίσιο της διαβούλευσης αλλά και στο πλαίσιο της συνάντησης του δικτύου δικαιοσύνης έδειξαν ότι τα κράτη-μέλη είναι μάλλον επιφυλακτικά όσον αφορά την κατάρτιση τέτοιων προδιαγράφων ποιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα, συμπέρασμά μας είναι ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να ε, υπάρξει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε οι εμπειρογνώμονες στο επίπεδο των κρατών μελών να εκπονήσουν οι ίδιοι κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και προδιαγραφές ποιότητας για την διαμεσολάβηση ε, στη βάση της οδηγίας ε, παρά λοιπόν το γεγονός ότι επί της αρχής το έργο αυτό θα πρέπει να έχει στο επίκεντρό του την αγορά, θα μπορούσε εφόσον ε, παραστεί ανάγκη να δοθεί και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Also rather controversial issue. Um, Ένα άλλο αμφιλεγόμενο ζήτημα και εδώ θα, ήθελα να ε, σας παραπέμψω και στα, στις απαντήσεις που λάβαμε στο πλαίσιο της διαβούλευσης αλλά και τις συζητήσεις που είχαμε με τα κράτη-μέλη ήταν ε, το ζήτημα της ε, υποχρεωτικής διαμεσολάβησης. Κάποιοι εμπλεκόμενοι φορείς συμπεραίνουν ότι η έλλειψη υποχρεωτικής δια, διαμεσολάβησης εμποδίζει την ε, επέκταση της ε, διαμεσολάβησης. Άλλοι λένε ότι από τη φύση της η διαμεσολάβηση πρέπει να έχει προαιρετικό χαρακτήρα γιατί ε, αλλιώς θα έχανε την ελκυστικότητά της ε, σε σχέση με τα δικαστήρια αν ε, καθίστατο υποχρεωτική. Ε, η θέση των κρατών μελών, όπως αποτυπώθηκε στις συνεδριάσεις του δικτύου, έδειξαν ότι τα κράτη-μέλη θα ήταν αρκετά επιφυλακτικά ως προς το να θεσπίσουν αλλαγές σε σχέση με, το, με τα όσα προβλέπει η οδηγία ως προς αυτό το θέμα. Το συμπέρασμα της ε, Κομισιόν λοιπόν είναι ότι το περιεχόμενο της ισχύουσας ε, οδηγίας και του άρθρου 5, παράγραφος 2, που, α, που ε, αφήνει αυτό το θέμα ε, στην αρμοδιότητα των κρατών μελών ε, είναι ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθεί και στο, στο μέλλον. Επίσης η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι η υποχρεωτική ε, διαμεσολάβηση μπορεί να επηρεάσει το δικαίωμα δίκαιης δίκης, πρόσβασης στη δικαιοσύνη, κάτι που κατοχυρώνεται ως δικαίωμα στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο θέμα που θέλω να αναδείξω είναι το ζήτημα της ε, εφαρμοσιμότητας, των, ε, της εκτελεστότητας των ε, αποτελεσμάτων της διαμοσολάβησης. Εδώ τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εμπλικόμενοι φορείς θεωρούν ότι η δυνατότητα εκτέλεσης των αποφάσεων της διαμοσολάβησης είναι πολύ υψηλές και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ πιθανό ότι εφόσον έχουν συγκαταθέσει στο να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση, τα, ε, ε, οι διάδικοι είναι τις περισσότερες φορές πιθανότατο να ακολουθήσουν τις ε, συστάσεις και, τις, α, α, τα αποτελέσματα της διαμεσολάβησης. Εδώ η Κομισιόν συμπεραίνει ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαμεσολάβησης θα μπορούσε ε, το ένα κράτος μέλος να ε, μπορεί να προβλέπεται να μπορεί να ζητήσει την, ε, να εκτελεστεί μια απόφαση της διαμεσολάβησης ακόμη και αν δεν υπάρχει συγκατάθεση του αντίδικου. Και τέλος θα ήθελα να φτάσω και στο τελικό συμπέρασμα βάσει των ε, στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας, φαίνεται ότι η εφαρμογή της οδηγίας ε, είχε σημαντικές ε, επιπτώσεις ως προς την νομοθεσία διαφόρων κρατών μελών. Όσον αφορά τις βασικές απαιτήσει για τη χρήση της διαμεσολάβησης σε διασυνολογικές υποθέσεις αστικές και εμπορικές, η οδηγία επίσης έδωσε κίνητρα ε, ώστε να ε, διαδοθεί η διαμεσολάβηση και σε εγχώριο επίπεδο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα κράτη-μέλη ε, διεύρυναν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και στις εγχώριες περιπτώσεις, υποθέσεις. Γι' αυτό η οδηγία έχει προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία καθώς ενίσχυσε την ευαισθητοποίηση, ενίσχυσε την ευαισθητοποίηση ε, είτε προκάλεσε τη δημιουργία είτε την ενίσχυση των προϋπαρχόντων συστημάτων διαμεσολάβησης. Επίσης, ε, όσον αφορά με βάση και το, το, το, το επίπεδο ε, που υπήρχε η διαμεσολάβηση, ο βαθμός στον οποίο υπήρχε η διαμεσολάβηση πριν από την θέσπιση αυτής της οδηγίας και τα προβλήματα που σχετίζονται με την λειτουργία των συστημάτων διαμεσολάβησης οφείλονται πολύ συχνά ε, στο γεγονός ότι υπάρχει χαμηλή ευαισθητοποίηση αλλά και ε, ελλειπής ε, εφαρμογή των κανόνων και των ελέγχων ποιότητας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει τροποποίηση της οδηγίας αλλά τόσο οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη μπορούν να ε, και πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για την περαιτέρω βελτίωση της ε, εφαρμογής. Τα κράτη-μέλη όπου δει θα πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειες προκειμένου να ενθαρρύνεται και να προωθείται η διαμεσολάβηση μέσω διαφόρων μηχανισμών όπως προβλέπει η οδηγία. Επίσης χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των υποθέσεων όπου τα δικαστήρια καλούν τα μέρη να χρησιμοποιήσουν τη μεσολάβηση για να φτάσουν σε συμβιβασμό. Εδώ η Κομισιόν έχει συντάξει και ένα κατάλογο βέλτιστων πρακτικών. Οι απαιτήσει ε, ε, ε, έχουν, έχουν υπάρξει προσπαθίες να υπάρξει υποχρεωτική αναφορά των διαδίκων στις προσφυγές τους στα δικαστήρια αν θα ήθελαν να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση και να ε, ενθαρρύνεται από την Κομισιόν να εξετάζεται η πιθανότητα χρήσης διαμεσολάβησης σε όλα τα ε, ε, επίπεδα. Η χρηματοδότηση, η οικονομικότητα μάλλον αυτών των, μορφών διαμεσολάβησης θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα κίνητρο που, για όλες τις πλευρές. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να συγχρηματοδοτεί έργα διαμεσολάβησης μέσω του προγράμματος Justice το οποίο είναι ανοιχτό προκειμένου να δίνεται χρηματοδότηση σε εμπλεκόμενους φορείς που ε, ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Επίσης, η Κομισιόν θα συνεχίσει να συμβουλεύει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαιοσύνης προκειμένου να δημιουργηθούν μεταξύ άλλων μια ε, ε, ισχυρότερη βάση δεδομένων σε σχέση με τη χρήση της διαμεσολάβησης. Επίσης ε, θα αξιοποιηθεί προς αυτό το σκοπό και η δυνατότητα που μας δίνει το Ευρωπαϊκό Πόρταλ για τη Δικαιοσύνη. Αυτά ήταν τα βασικότερα στοιχεία της έκθεσής μας. Νομίζω ότι μπορούν αυτά που σας είπα να αποτελέσουν και μια καλή βάση για την συζήτηση που θα έχουμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάιμπαχ και τώρα να καλωσορίσω τον καθηγητή Τζουζέπε Ντεπάλο ο οποίος ε, είναι υπεύθυνος για επίλυση διαφορών και ειδικό για το θέμα αυτό στην νομική του Μίτσελ Χάμιλαϊν. Καθηγητά Ντεπάλο, έχετε 10 λεπτά για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Έχω κάποια πράγματα και εγώ να πω σήμερα. Κυρίω γιατί ο τίτλο ε, τη παρουσίας όπω τον βλέπετε στην οθόνη, έχει ένα λάθο στην δεύτερη γραμμή. Θέλουμε μια πιο ισορροπημένη σχέση μεταξύ τη διαμεσολάβηση και των ε, δικαστικών ε, διαδικασιών. Η οδηγία του 2008 είναι πραγματικά ένα ορόσημο στην, στο ολονομικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία έχει σαρώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Όμω οι πραγματικοί στόχοι τη οδηγία πόρο απέχουν από την επίτευξή του. Πραγματικά αυτό που θέλαμε ήταν περισσότεροι, σε περισσότερες εταιρείε να χρησιμοποιούν τη διατησία για να ε, επιλύσουν διαφορές. Όμως, τα δεδομένα δείχνουν ότι για κάθε 100 υποθέσεις που εκδικάζονται, είναι λιγότερο από μία σε περιπτώσεις της ε, διαιτησίας. Το 1 προς 100 δεν είναι καλή σχέση. Το 2014 η μελέτη για την ανανέωση του όλου θέματος, την αναθέρμανση της εξέτασής του, έδειξε ότι υπάρχουν θέματα ποιότητας, εμπιστευτικότητας και επιβολής της οδηγίας. Αυτά τα τρία στοιχεία οδήγησαν στην ε, διάθεση να αναθεωρηθεί αυτή η οδηγία. Το στοιχείο που θα μπορούσε να αυξήσει τον αριθμό των υποθέσεων ε, διαιτησίας υπάρχει ήδη στην οδηγία, το άρθρο 5.2 που το βλέπετε τώρα και στην οθόνη. Εκεί η εθνική νομοθεσία θα μπορούσε να απαιτεί τη χρήση διατησίας εφόσον διαφυλάσσεται το δικαίωμα των αντιδίκων ε, να ε, προσφύγουν στα δικαστήρια. Τώρα, στην Ιταλία 8% αστικών και πενικών υποθέσεων πρέπει οπωσδήποτε να περάσουν από την περίπτωση της διαιτησίας. Δηλαδή 200.000 διαιτησίες ε, αναμένονται ετησίως 20 φορές παραπάνω από σε οποιοδήποτε άλλο κάτω μέλος. Πριν από 6 χρόνια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διευκρίνησε πώς μπορεί να γίνει η απέτηση για τη διατησία ε, συμβατή με το δικαίωμα πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Πρέπει λοιπόν να μην είναι δεσμευτική, να είναι γοργή η εκδίκαση και να είναι ε, χαμηλό το κόστος της διατησίας. Αυτή τη στιγμή Πρέπει να απαιτείται η προσπάθεια για την ε, προσφυγή σε διατησία, αν θέλουμε το δικαστικό σύστημα να αποτελεσματικότερα. Σήμερα, όλο ένα και, και μεγαλύτερο αριθμό χωρών απαιτούν κάποιε προσπάθειες διατησία πριν ξεκινήσει η διαδικασία αυτή καθεαυτή. Η μελέτη της Επιτροπής συστήνει και παραθέτω εδώ να υπάρχει μια ε, προκαταρκτική δικαστική υπόθεση όπου, ένας αποφασίζει από την το κατά πόσο η διαφορά μπορεί να επιληθεί καλύτερα στα πλαίσια της ειδησία παρά με δικαστική διαδικασία. Αυτή η επιλογή, εφόσον σωστά διακρίνει μεταξύ της υποχρεώσης των μερών να συναντηθούν με ένα διαιτητή τουλάχιστον μία φορά, κάτι που είναι απολύτως θεμητό, και την υποχρέωση να επιληθεί διαφορά μέσω διατησία, που θα ήταν πραγματικά παραβίαση του άρθρου 47, αυτά τα δύο μπορούν να συνδυαστούν και να βρεθεί μια μέση οδό. Επίση, η αποτέμιση του κατά πόσον η διατησία μπορεί να επιλύσει μια συγκεκριμένη υπόθεση ή όχι, είναι κάτι που το κάνουν καλύτερα οι αντίδικοι με του διαιτητέ του μαζί στη διαδικασία τη διαιτησία αυτή καθεαυτή. Όχι ξεχωριστά σε μια ενημερωτική συνεδρία διατησία, όπου μετά μπορεί να να ακολουθηθεί από απόπειρα να ξεκινήσει η διαδικασία διευθυνσία. Έτσι, αυτή η, αυτό το φιλτράρισμα της διευθυνσία θα μπορούσε να είναι μια εύφυης λύση μεταξύ δύο αρχών. Από τη μια την απολύτη ελευθερία των μερών, αν θέλουν να ε, επιλύσουν ή τη διαφορά τους, και από την άλλη την αποδεδειγμένη ανάγκη να απαιτηθούν σοβαρές προσπάθειες διευθυνσίας. Κάποιοι θεωρούν ότι οι αντίδικοι, τα μέρη δηλαδή, αν απευθυνθούν στους διαιτητές, θα, θα βρουν αντίσταση από τους δικηγόρους. Πριν από πέντε χρόνια στην Ιταλία έγινε απεργία, όντως. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν αφισβητεί όμως τη διαιτησία. Μάλιστα, πριν από ένα τρίμηνο, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Ιταλίας, ετήσιο, στο ετήσιο συνεδριό του, υπερψήφισε τις ε, ε, ε, πρωτοβουλίε για διαιτησία και ζητήθηκε το πεδίο της διαιτησία να επεκταθεί. Δεν υπάρχει βεβαίω εγγύηση ότι η ίδια μεταβολή θα γίνει και σε άλλες χώρες όπου η διαιτησία θα απαιτηθεί και ε, θα χρησιμοποιείται σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Όμως η Ιταλία δεν είναι η πρώτη χώρα όπου οι δικηγόροι πρώτα είναι πρώτοι πολέμοι και μετά είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του όλου συστήματος της αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει αρκετή κουλτούρα υπέρ τη διαιτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί επιχειρηματολογούν ότι ο λόγο που δεν χρησιμοποιείται αρκετά η διαιτησία είναι γιατί δεν την γνωρίζει ο κόσμο. Χρειάζονται επενδύσει στην ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση προκειμένου να υπάρξουν περισσότερε περιπτώσει διαιτησία. Βεβαίω, ε, η στάση που θα είναι υποφελή για την κοινωνία, δηλαδή λύση με διαιτησία για πολλέ περιπτώσει, είναι η ποιότητα και είναι σημαντικό να υπάρχουν κίνητρα, εκπαιδευτικές ευκαιρίες και αυτά θα ε, επιτρέψουν να αναπτυχθεί περισσότερο το σύστημα διατησίας αφού αποφασίσει ο νομοθετής. Ο νομοθέτης. Ε, το να προστρέξει κανείς ή όχι στη διευθυνσία έχει και ιδιωτικές και δημόσιες συνέπειες, διότι αυτή τη στιγμή οι αντιδικοί πληρώνουν μόνο το 24% του συνολικού, ε, της συνολικής δικαστικής διαδικασίας. Οι περισσότεροι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τη δικαστική αλλογή, αλλά ε, πρέπει να χρησιμοποιούνται συνετά οι πόροι αυτοί για την δημόσια και είναι και περιορισμένοι. Μια χρήσιμη απεικόνηση της ε, σχέσης μεταξύ της νομοθετικής διαδικασίας και της κουλτούρας προέρχεται από την ευρωπαϊκή χώρα με τις περισσότερες διαιτησίες τώρα. 81,1% στην Ιταλία είναι υποχρεωτικές ε, διαιτησίες. 8,3% είναι οι εθελοντικές. Και αυτές οι εθελοντικές δεν υπήρχαν πριν την απέτηση. Άρα η πράξη βλέπουμε ότι καλλιεργεί με τη σειρά της την ε, όλη κουλτούρα υπερτιδιατησίας η οποία ξεκινά όντω από την νομοθετική και την νομική υποχρέωση, όπω δείχνουν οι στατιστικέ ε, στην Ευρώπη και αλλού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, φαίνεται να έχει δύο βασικέ επιλογέ για να ενθαρρύνει τη χρήση τη διαιτησία και να φέρει την ισόρροπη σχέση μεταξύ ε, και και εκδίκασες υποθέσεων. Πρώτα απ' όλα να αλλάξει το άρθρο 5.2 ε, της οδηγίας και να αλλάξει και αυτό το πρώτερο φιλτράρισμα που προβλέπετε. Δηλαδή τα μέρη θα πρέπει έστω με μία αρχική ε, συνεδρία διατησίας να ενημερωθούν και μετά εθελοντικά να περάσουν ε, σε πραγματική διατησία. Έτσι θα υπάρχει και ε, πλήρης ελευθερία και αποτελεσματικότητα. Η δεύτερη επιλογή είναι να βελτιωθεί η χρήση του σημερινού άρθρου 52. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εφόσον οι ελευθερινοί στόχοι τη οδηγία δεν έχουν ε, ε, επιτευχθεί εδώ και 10 χρόνια, ο νομοθέτης έχει περισσότερο απονομική υποχρέωση να κάνει κάτι γι' αυτό. Τον Δεκέμβριο του 2014 η Επίτροπος Γιούροβα χαρακτήρισε εντυπωσιακά τα αποτελέσματα της μελέτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ονομάστηκε rebooting. Εδώ μας ενδιαφέρει να βρούμε μια σωστή λύση μεταξύ διαμεσολάβησης και διαιτησίας. Μάλλον ε, και εκδίκασης των υποθέσεων με δικαστικές διαδικασίες. Θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε δις ευρώ και εκατομμύρια ημέρες από ε, περιτές εκδικάσεις υποθέσεων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν φαίνεται να ε, καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσματα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει συνένεση και πολλές δυνατότητες με εύλογες προσπάθειες υπέρ της Διευθυνσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να περάσουμε σε κάτι καλύτερο, ακολουθώντας αυτές τις συστάσεις. Αν γίνει αυτό, σε ένα χρόνο από τώρα, ίσως και σε αυτή την ίδια την αίθουσα, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να μετράμε και να γιορτάζουμε για τον οικονομικό και κοινωνικό θετικό αντίκτυπο τη χρήση της Διευθυνσία και εκ μέρου του κυρίου Ντούρσο, αλλά και την ομάδα των εμπειρογνωμόνων που με βοήθησαν στην εκπόνηση τη έκθεση αυτή. Βλέπετε τα ονόματα του στην οθόνη. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Εκτός μικροφώνου ο μιλητή. now... Προχωρούμε τώρα με την παρέμβαση του δικαστή Τζέφρι Βόσο από το Αντώτατο Δικαστήριο. Θα μας μιλήσει για τη σχέση μεταξύ της επίσημης και της ανεπίσημης δικαιοσύνης, αντικείμενο μια συνεχούς διαδικασίας που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2016. Λόρδα, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Ε, θα παρατηρήσατε ότι έχω λίγο βήχα και αν καταρρεύσω κάποια στιγμή στο πάτωμα, να ξέρετε ότι δεν είναι σκεμμένο, να με συγχωρέσετε. Το κοινό εγχείρημα για το οποίο θα, ήθελα να σας μιλήσω μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικτύου ε, Συμβούλων για το Δικαστικό Σκέλος και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου ε, δημιουργήθηκε λοιπόν αυτή η διαδικασία διότι έχουμε εκθετικά, εκθετική αύξηση διαφόρων μορφών επίλυσης διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκθετική αύξηση διαφόρων εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών. Έχουν προκύψει προβλήματα από δικαστικής πλευράς, αφέστατα. Και τα αναγνωρίσαμε αυτά και αποφασίσαμε ότι τρεις είναι οι πιθανές εκδοχές που μπορούν να προκύψουν από αυτό το κοινό εγχείρημα, το οποίο καλεί ε, να συμβάλλει το δικαστικό σκέλος, ο πανεπιστημιακός κλάδος, αλλά και οι δικηγόροι, το νομικό επάγγελμα. Θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια δήλωση ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών σύμφωνα με την προσέγγιση που θα έπρεπε να υιοθετήσουν τα δικαστήρια και οι δικαστές όταν καλούνται να αλληλεπιδράσουν με όλα τα ίδια εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών. Και άρα θα υπήρχαν κατευθυντηρίες γραμμές για τα προκαταρκτικά, για τις διαδικασίες που θα πρέπει να υιοθετηθούν όταν έχουμε εναλλακτική επίλυση διαφορών και όταν ε, ένα δικαστήριο καλείται να τοποθετηθεί επί της εναλλακτική επίλυση διαφορών ή της διαμεσολάβησης και άρα να μειωθεί η προσφυγή στους, στο δικαστήριο. Δεύτερη πιθανή έκβαση ήταν να υπήρχε αντίστοιχη δήλωση με αυτή των ευρωπαϊκών των πρακτικών, αλλά κυρίως να δοθεί έμφαση στο πώς όσοι καθορίζουν και καθοδηγούν το μηχανισμό επίλυσης διαφορών τον εναλλακτικό, πώς θα πρέπει αυτοί να λιλεπιδρούν και να συνεργάζονται με τα δικαστήρια και τους δικαστές. Και πάλι στόχος θα ήταν να μειωθεί ο κίνδυνος αδικιών από αυτούς τους εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Και τρίτη έκβαση ήταν να γίνουν συστάσεις για το καλύτερο ευρωπαϊκό μοντέλο που θα μπορούσε να καταρτιστεί και να υπάρξει για να υπάρχει πρόσβαση με συνέπεια ε, σε αυτούς τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών ε, για διαφορά αιτικά είδη διαφορών και για τους τρόπους με τους οποίους θέλουν τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν. Δεν θα πω πολλά λόγια γι' αυτό. Είναι όμως εξαιρετικά σημαντικό, γιατί εκεί όπου υπάρχουν διαφορετικές εναλλακτικές διαθέσιμες, εναλλακτικές διαθέσιμες ε, λειτουργίες σε μηχανισμού επίλυσης διαφορών, ο καταναλωτής δικαστικών υπηρεσιών πρέπει να ξέρει πού θα τις βρει και πώς θα έχει πρόσβαση σε αυτές. Δεν έχει γίνει Πολύ δουλειά σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές, για τους δικαστές όταν αντιμετωπίζουν εναλλακτική επίλυση διαφορών, ούτε αντιστρόφους. Και εγώ προεδρεύω μια ομάδα η οποία ανησυχεί ιδιαίτερως για τις ευπαθείς ομάδες, για τα ευπαθή αν θέλετε ε, διάδικα μέρη, τις μικρές επιχειρήσεις, τις οικογένειες, τα άτομα που συχνά νιώθουν πίεση να συνενέσουν να υπάρξει μηχανισμός επίλυσης διαφορών εναλλακτικός και να υπάρξει διαμεσολάβηση χωρίς να κατανοούν απολύτως τα νομικά τους δικαιώματα. Τίποτα από αυτά που λέω δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως τίποτα άλλο παρά μόνο η ολόθερμη στήριξη στην αυξημένη χρήση της διαμεσολάβησης και της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και γενικότερα και ειδικότερα. Ωστόσο πρέπει να επαγρυπνούμε έναντι των κινδύνων που ε, γεννά η εναλλακτική επίλυση διαφορών εάν γίνει εσφαλμένη χρήση αυτής. Δεν θέλω να ε, καταχραστώ του χρόνου σας και από τη στιγμή που δεν έχω καταρρεύσει με παροξυσμικό βήχα σημαίνει ότι πάνε καλά τα πράγματα προς το παρόν και γι' αυτό μπορώ εν συντομία να προχωρήσω ε, λέγοντας τα εξής. Πρώτον, ο κίνδυνος να να υπάρξει άρνηση για ανεξάρτητο δικαστικό προσδιορισμό έναντι του ατόμου. Δηλαδή, μεγάλοι κρατικοί οργανισμοί, μεγάλες επιχειρήσεις μπορεί να προωθήσουν την εναλλακτική επίλυση διαφορών και οι πολίτες να νιώθουν ότι απαιτείται να συνενέσουν στην επίλυση, στη ρύθμιση, την εξοδικαστική αν θέλετε. Ενώ το άρθρο 9 ε, ε, λέει ρητά ότι πρέπει τα διάδικα μέρη να ενημερωθούν ότι δεν υποχρεούνται να συνενέσουν και θα πρέπει να ε, γίνει αυτό αντιληπτό. Ποια είναι η βέλτιστη πρακτική που θα πρέπει να υιοθετήσουν οι οι δικαστικές αρχές. Σίγουρα οι δικαστικές αρχές θέλουν να μειωθεί ο φόρτος εργασίας των δικαστηρίων. Ως εκ τούτου, ορισμένες δικαστικές αρχές θεωρούν ότι αξίζει τον κόπο ο κίνδυνος κάποιες διαφορές να ρυθμιστούν με έναν εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών και ας μην υπάρχουν όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες για την ασφάλεια δικαίου και την ε, για ε, ε, τη Βουλή στη συνένεση των διαδίκων μερών. Σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο να κάθε πολίτης να δέχεται νομική συμβουλή, ανεξάρτητη νομική συμβουλή για οποιοδήποτε ζήτημα. Μπορεί ο πολίτης να μην ζητήσει σύμβουλη, γιατί θεωρεί ότι η διαφορά είναι ίσονος σημασίας. Μπορεί να λάβει ε, την ορθολογική απόφαση να γλιτώσει χρόνο και χρήματα και να, γι' αυτό να μην έχει νομική σύμβουλη. Ή μπορεί να είναι ο ίδιος σε θέση να αξιολογήσει τους νομικούς κινδύνους από την άγουσα που ε, επιλέγει. Η σύγχρονη διαδικτυακή λειτουργία επίλυσης διαφορών, ο ιδιο σε θεση να αξιολογησει τους νομικους κινδυνους απο την αυτός ο διαδικτυακός έχει σχεδιαστεί με σκοπό να αποκλείσει από αυτή τη διαδικασία τους νομικούς εκπροσώπους. Επομένως υπάρχει ενδεχομένως ε, βαρός κίνδυνος ότι ε, πολίτες θα συμβιβαστούν για πάρα πολύ λίγα γιατί δεν γνωρίζουν τι αξίζει η απέτησή τους. Και αυτό ισχύει στις οικογενειακές υποθέσεις όπου τα συναισθήματα είναι έντονα και η επιθυμία να συμβιβαστεί κανείς θεωρείται επίγουσα ε, επιθυμία για διάφορους άλλους λόγους που δεν έχουν σχέση όμως με την ένομη τάξη. Και σε άλλα πεδία το βλέπουμε αυτό. Κάθε φορά που προτείνεται ένας εναλλακτικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών, όποιος και να το προτείνει, δικαστής ή άλλος, θα πρέπει να διασφαλιστεί και να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ότι δεν ε, γίνεται επίκληση αυτής της διαδικασίας για να αποφύγει κανείς τις νομικές του υποχρεώσεις και θα πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες που να διασφαλίζουν ότι είναι ένα παιχνίδι επίσης όρης και για τα πιο ευπαθή διάδικα μέρη οι διαμεσολαβητές και οι όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις ενδεχομένω δεν είναι σωστά καταρτισμένοι. Και αυτό είναι το τρίτο θέμα που θα ήθελα να δείξω Και τέταρτο θέμα είναι ο κίνδυνος τα διάδικα μέρη να μην γνωρίζουν και να μην κατανοούν ε, απολύτως τις διαθέσιμες μεθόδους και μίλησα γι' αυτό προηγουμένως. Ουσιαστικά είναι ένα αρκοπέδιο για τον ατομικό καταναλωτή δικαστικών υπηρεσιών να ξέρει πώς μπορεί να ρυθμίσει τις διαφορές του με μια εταιρεία κοινή ωφελία, με μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών, με τον οποιοδήποτε τρίτο που έχει ε, θεσμοθετήσει μια διαδικασία διαμεσολάβησης, κάτι που ισχύει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέμπτον, υπάρχει κίνδυνος από έναν που λαμβάνει τις αποφάσεις και δεν είναι αναγνωρίσιμος και βρίσκεται στο διαδίκτυο. Έχουμε το σύστημα στο eBay, το οποίο επιλύει κυβερνητικές ε, διενέξεις, δηλαδή διαφορές και διενέξεις στον κυβερνοχώρο και μάλιστα περηφανεύεται ότι επιλύει περισσότερες διενέξεις από ό,τι τα ίδια τα δικαστήρια, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί τελικά. Και επειδή υπάρχει εθελούσια επιλογή και επειδή δεν υπάρχουν τα απαραίτητα προσόντα, μπορεί να μην χρησιμοποιηθούν επαρκώς. Και οι δύο προηγούμενοι ομιλητές αναφερθήκαν ήδη για το, στο θέμα αυτό. Και τέλος, κάτι που υπάρχει ως κίνδυνος και τον υποτιμούμε είναι οι καταχρήσεις από πλευράς μεγάλων κρατικών ή εμπορικών ε, οντοτήτων και φορέων που επιβάλλουν τη βούλησή τους στους καταναλωτές κάθε φορά που οι τελευταίοι έχουν διαφορά με μεγαλύτερη οντότητα, με κάποιο μεγαλύτερο φορέα. Αυτός ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αξιολογηθεί και να εκτιμηθεί και είναι υπερβολικά σημαντικό να μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτούς τους κινδύνους. Αυτό το προσπαθούμε στη, στο δικό μας έργο, δηλώνουμε τις βέλτιστες πρακτικές και ελπίζω να συμβάλλουμε στην καλύτερη διαμεσολάβηση και πρακτική εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Και τώρα ο, ο κύριος Φέλξ Στέφεκ, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, που θα επικεντρωθεί στην, ε, στο, στη σχέση μεταξύ της οδηγίας για τη μεσολάβηση και τον κοινωνισμό για τις online διαφορές, να εντοπίσει τις διαφορές και να μας παρουσιάσει το νομικό πλαίσιο. Έχετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή και τον Πρόεδρο για την πρόσκληση που με απίφθηνε να μιλήσω για αυτή τη σχέση, για τη σχέση μεταξύ της διαμεσολάβησης και άλλων μορφών αλλακτική επίλυσης διαφορών. Θα ήθελα να κάνω τρία σχόλια. Πρώτον, θα ήθελα να σχολιάσω την πρόοδο και τις ελλείψεις που ε, ε διαπιστώθηκαν με βάση τα τρία ε, νομοθετικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Επίσης, θα ήθελα να παρουσιάσω μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την αναρτική επίλυση διαφορών, να παρουσιάσω μέσα και εργαλεία για τη βελτίωση της εναλλακτική επίλυσης διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτον, ποια θα μπορούσε να είναι το μέλλον. Ποιο θα μπορούσε να είναι το μέλλον. Θα ήθελα να προτείνω τρεις ε, δρόμους ε, δράση. Πρώτον, όσον αφορά τις ε, εξειδικευμένες μορφές εναλλακτικής επίλυση διαφορών τα βασικότερα εργαλεία και ιδίω η οδηγία έχει βελτιώσει την κατάσταση γύρω από την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Ωστόσο, μία μορφή από αυτές τις εναλλακτικέ επιλύσεις διαφορών καλύπτεται από τον νόμο και αυτή είναι η διαμεσολάβηση. Η οδηγία ADR και ODR ε, προσεγγίζουν με γενικό τρόπο την διαμεσολάβηση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο μέσο για εσωτερικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών, συμβιβασμού, διακανονισμού, ούτε ε, διαδικασίες ε, ουδέτερων αξιολογήσεων, δεν υπάρχουν συστήματα διαμεσολάβησης, ε, διαιτησίας ή δικαστικών προτάσεων και πολλές άλλες εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών που υπάρχουν. Συμπεραίνω ότι αυτή τη στιγμή οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά από διάφορες μορφές εναλλακτικής επίληξης διαφορών που να ε, εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα ποιότητας. Δεύτερον, ελλείψεις και προβλήματα σε, σε σχέση με, την με τη, όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των διαφόρων μαρφών. Τα, τα νομοθετικά εργαλεία ασχολούνται μόνο με τη σχέση μεταξύ διαμεσολάβησης και δικαστηρίων και όχι μεταξύ ε, επιμέρους εναλλακτικών μορφών επίλυση διαφορών. Υπάρχουν κανόνες όσον αφορά την ε, εμπιστευτικότητα της διαμεσολάβησης σε δικαστικές διαδικασίες και όσον αφορά το κόστος. Τέτοιοι κανόνες ε, χαρακτηρίζονται από ποιότητα και από διαφάνεια ε, ιδίως όταν προηγείται μια... Ε, αν όμω εξετάσει κανείς αν υπάρχει ε, καλή εφαρμογή αυτής της διαμεσολάβησης, η απάντηση είναι αρνητική. Ε, άρα οι πολίτες ε, ε, είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουν μία και μόνο μορφή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Τρίτον, πρόοδος και ελλείψεις όσον αφορά τις ε, βασικές αρχές του κανονισμού. Θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαία αντίληψη για τη ρύθμιση του, της διαμεσολάβησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω κανονισμού. Θα απαιτούνταν για κάτι τέτοιο μια συναντήληψη όσον αφορά ε, τον, τον, μια κοινή αντίληψη των ε, μορφών αυτής της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και ε, πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αυτές σε διασυνορικές υποθέσεις. Θα ήθελα να σας υποβάλω σε μια δοκιμή. Να σας ρωτήσω αν υπάρχει μία και ενιαία ε, βασική αρχή όσον αφορά το κόστος των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών. Γνωρίζετε δηλαδή ε, όσον αφορά το κόστος ε, των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών, διαιτησία, διαμεσολάβηση κτλ. Αν εσείς ή ε, το διάδικο μέρος ή το κράτος θα βαρύνεται με το κόστος αυτής της διαδικασίας. Θα ήθελα να πω ότι εφόσον δεν υπάρχει μια τέτοια επί της αρχής προσέγγισης, οι πολίτες πολλές φορές επιλέγουν εκείνη την εναλλακτική μορφή επίλυσης διαφορών που δεν υπηρετεί τα συμφέροντά τους. Και θα ήθελα να πω σε σχέση με την έκθεση της Επιτροπής ότι το έλλειμμα όσον αφορά την ε, επιλογή του σωστού τύπου διαμεσολάβησης ή εναλλακτική επίλυση διαφορών δεν ε, οφείλονται στις ελλείψεις της, ε, της ε, οδηγίας ε, για τη διαμεσολάβηση, αλλά όλων των νόμων που σχετίζονται με τι αναλλακτικέ μορφέ επιλογή διαφορών. Πώ θα μπορούσε λοιπόν να. Ε, τι μορφή θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο ένας τέτοιος νόμος. Πρώτον, χρειαζόμαστε μια εύρυθμη ε, λειτουργία και ένα εύρυθμο πλαίσιο λειτουργίες Αυτό δεν θα πρέπει να αφορά μόνο με τις νομικές τυπικότητες, αλλά την εφαρμογή στην πράξη. Τα διάδικα μέρη μπορούν ε, να διακριθούν ε, σε ε, συγκεκριμένες κατηγορίες. Πρώτον, ε, έλεγχος της συγκατάθεσης, αν τα μέρη συμφωνούν. Προ, έλεγχος διαδικασίας, έλεγχος των αποτελεσμάτων της διαδικασίας, της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας, όπου χρειάζεται ε, συγκατάθεση για τη δεσμευτικότητα των αποτελέσματων. Ε, ουδετερότητα και έλεγχος της ε, πληροφόρησης που αφορά ε, την ιδιωτικότητα των πληροφοριών που συλλέγονται στη διαδικασία. Δεύτερον, χρειάζεται επιλογή πολιτικής. Εδώ τα, οι πολίτες αλλά και οι αρχές θα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο αυτής της ε, διαδικασίας. Και αυτό συμβαδίζει πλήρως με την ε, χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ θέτω δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ε, το άτομο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της. Το ότι οι διαφορετικές υποθέσεις απαιτούν διαφορετικές μορφές αναρακτικής επίλυσης διαφορών μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε διαφορετικές μορφές αναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Και τρίτον, όσον αφορά την επί της αρχής ρύθμιση, ε, υπάρχουν ε, τέτοιες και στον ίδιο τον κανονισμό. Αυτές οι αρχές θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις μορφές αναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Ε, είχα τη χαρά μαζί με 16 συναδέλφους να κατακτήσουμε έναν οδηγό ε, για αυτήν την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα όσον αφορά τα, τα προσόντα. Λέει ότι όσο λιγότερο ε, τα μέρη ε, ελέγχουν την, τη σύνθεση ή τα προσόντα του διαμεσολαβητή, τόσο περισσότερο το κράτος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ουδετερότητά του. Αυτό αντικατοπτρίζει και τη συζήτηση που σχετίζεται με, την, με τα προσόντα των διατητών, των διαμεσολαβητών, των ε, συνηγόρων και ε, είναι προφανές ότι τα ζητήματα αυτά χρειάζονται περισσότερη δουλειά. Χρειάζεται να εξασφαλιστεί η αυτονομία και η προστασία των επαγγελματιών του χώρου έναντι μη καταρτισμένων προσώπων. Αυτή η αρχή σχετίζεται με την εύρυθμη λειτουργία των μηχανισμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Τα χαρακτηριστικά που ε, περιέγραψα για τους διαμεσολαβητές είναι ο έλεγχος της ενεργοποίησης, του, των αποτελεσμάτων και κυρίως την επιρροή των μερών όσον αφορά την επιλογή του διαμεσοβαλαβητή. Πώς αυτό μπορεί να μετουσιωθεί σε πρακτικά βήματα. Πρώτον, θα ήθελα να προτείνω να, ε, ότι χρειάζονται περισσότερα ε, εργαλεία εναλλακτική επίλυση διαφορών. Κάτι που θα ε, άρει και την ανισορροπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή τα περαιτέρω ε, εργαλεία εναλλακτική επίλυση διαφορών θα μπορούσαν να μοιάζουν με τη διαμεσολάβηση ε, όπως είναι οι διαδικασίες διαμεσολαβητών ή οι γνωμοδοτήσεις ε, εμπειρογνωμόνων σε περιπτώσεις διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων. Στο επίπεδο κράτος μέλος θα μπορούσαν τα αστικά δικαστήρια να μετατραπούν σε δικαστήρια διαμεσολάβησης χρειάζεται να ε, ξεκαθαριστεί η συγκεχημένη σχέση μεταξύ των διαφόρων μορφών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Ένα οριζόντιο εργαλείο μπορεί να ασχοληθεί με όλα αυτά τα ζητήματα ή θα μπορούσε να ενταχθεί σε συγκεκριμένα εργαλεία εναλλακτική επίλυση διαφορών. Και τέλος θα ήθελα να προτείνω ένα εργαλείο ε, μηχανισμού που θα μπορούσε να άρει την ε, έλλειψη μιας επί της αρχής προσέγγισης επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μπορούσε να εξασφαλίσει την συνεκτικότητα ε, μεταξύ των διαφόρων μορφών επίλυσης, εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αλλά και σε διασυνοριακό πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο αναφοράς θα μπορούσε να βασίζεται στο λειτουργικό πλαίσιο αναφοράς, στις ε, επιλογές πολιτικές, ε, πολιτικής που μόλις σας παρουσίασα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν μια αξιοσημείωτη πρωτοβουλία και θα ε, αποτελούσε μια σημαντική βελτίωση όσον αφορά την ισχύουσα κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία σας και τώρα να ξεκινήσω τη συζήτηση για ζητήματα που ήδη έχουν θυγεί και να δώσω στους συναδέλφους το λόγο για να θέσουν ερωτήματα και να έχουμε απαντήσει από τους ομιλητές μας. Ο κύριος Ντεπίντο έχει πει ότι μπορεί να θέσει ερωτήσεις. Ήθελα να θέσω μια ερώτηση. Ε, αλλά περισσότερο από ερώτηση, κάποιες παρατηρήσεις ήθελα να κάνω σε σχέση με την διαδικασία της διαιτησίας και την όλη πολιτική περί που ακολουθούν κάποιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ξεκινήσω με μία ερώτηση. Γιατί η διαιτησία, μάλλον τι προσφέρει η διαιτησία, τι το θετικό, που η δικαιοσύνη των δικαστηρίων, η συμβατική, δεν μπορεί να το προσφέρει. Η απάντηση ως τώρα είναι ότι η διαιτησία είναι πιο γοργή, πιο ανεπίσημη και πιο κοντά στους ίδιους τους πολίτες και πιο φτηνή. Εγώ απαντάω με μια αντερώτηση. Γιατί τότε να μην γίνουν μεταρρυθμίσει ώστε να επιστρέψει η δικαιοσύνη όπω παρέχεται στα δικαστηρία και να γίνει πιο ανεπίσημη, πιο φτηνή, πιο γοργή και πιο κοντά στου πολίτε. Αντί να επαναλαμβάνονται υπηρεσίε, να γίνει μια μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματο, του ίδιου του οικοδομήματο τη δικαιοσύνη και να παρέχεται από εκεί το ίδιο πράγμα. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει μια διπλή απώλεια. Απώλεια χρήματος και απώλεια χρόνου. Διότι στην πράξη τα άτομα, ε, οι άνθρωποι όταν πηγαίνουν ε, για επίλυση μιας διαφοράς τους ενδιαφέρει κάποιος ε, που είναι εκτός της διαφοράς να λάβει ακριβώς μία τέτοια απόφαση ουδέτερη. Δηλαδή πηγαίνουν στο δικαστήριο, στο το δικαστήριο με την κυρίαρχη ε, απόφασή του να επιλύσει το ζήτημα. Τα δικαστήρια φαίνεται ότι έχουν εξαντλήσει τις διαμεσολαβητικές τους ε, και διαιτητικές τους δυνατότητες. Αυτές μπορεί να επιτρέψει η εκδίκαση μιας υπόθεσης. Τέλος, ε, πρέπει να πω τα ωφέλη της διαιτησίας είναι προφανή. Και υπάρχουν ε, κάποιες ε, πτυχές όμως που δεν είναι και τόσο προφανείς και το θέμα είναι ότι πολλές φορές οι διάδικοι εμφανίζονται ενώπιον του δικαστή χωρίς να καταλαβαίνουν πώ ακριβώ μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά του, χωρί να καταλαβαίνουν νομικώ τι ακριβώ διακυβεύεται. Ο δικαστή, ένα κράτο δικαίου, δεν είναι ο βασιλιά Σολομώντα που αποφασίζει ξαφνικά με τη θεία φώτιση και με μια ανώτερη νόηση που είναι υπερφυσική πώ θα αποφασίσει. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία στη διάθεση του δικαστή και τα συγκεκριμένα στοιχεία των διαδίκων. Η δικαιοσύνη είναι επίσημη ακριβώς και είναι επίσημο το σύστημα αυτό, διότι το, η ίδια επισημότητα του συστήματος εξασφαλίζει τους πολίτες κατά της αυθαιρεσίας. Λεγόταν το 19ο αιώνα ότι ακριβώς ε, η επίσημος χαρακτήρας, τυπικότητα του δικαστικού συστήματος εξασφαλίζει από την αυθαιρεσία. Πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε κατά πόσον τα κράτη ε, είναι λογικό να προωθούν εναλλακτικέ μορφέ απόδοση δικαιοσύνη από την ίδια τη δική του τη δικαιοσύνη. Είναι προφανέ. Ε, αλλά πώ ε, τα κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βλέπουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταργείται ίδια στα δικαστήρια υπέρ δικαστηρίων δικαστηρίων πιο αυθαίρετων ε, που να υπόκεινται στους κανόνες του διεθνούς εμπορίου που να ε, υποκλέπτουν ουσιαστικά την κυριαρχία από το ίδιο το δικαστικό σύστημα και από τα ίδια τεχνικά κράτη και να παρέχεται δικαιοσύνη από διαιτητές, από πρόσωπα τα οποία ορίζονται αυθρέτως από τα, τους διαδίκους. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι δημόσια, ώστε κανείς να μην μπορεί να την αποδώσει εμέσως ή αμέσως. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι δημόσια, να έχει δημόσιο πρόσωπο. Και για να έχει δημόσιο πρόσωπο Μάλλον, εφόσον έχει δημόσιο πρόσωπο, τότε μόνο είναι μέρος της εθνικής κυριαρχίας των κρατών. Ε, κάτι που είναι ε, της στόχος, δηλαδή να είναι αμερόληπτη και ουδέτερη. Οι δικαστές ε, είναι, έχουν μπροστά τους τους διαδίκους ε, και οικονομικά αλλά και πολιτιστικά είναι πολύ περισσότερο προστατευμένοι πολίτες ενώπιον αυτών των δικαστών παρά έναντι των διαιτητών. Πρέπει λοιπόν να ε, σκεφτούμε κατά πόσον οι διάδικοι στην πραγματικότητα, στην πράξη, προστατεύονται περισσότερο ενώπιον ενό δικαστή ή ενό διαιτητή. Πώ λοιπόν τα κράτη να παρέχουν εναλλακτικέ στο ίδιο του το δικαστικό το σύστημα, χωρί να έχουν επιχειρήσει καν τι ε, μεταρρυθμίσει που απαιτεί το δικαστικό σύστημα το ίδιο. Πρόεδρε, και θα ολοκληρώσω, μια εικόνα που χρησιμοποιείται πολύ στη χώρα μου για τη δικαιοσύνη είναι η εξή. Εάν ένα πολίτη από τη Γαλλική Επανάσταση λόγου χάρη. Κάποια στιγμή έμενε άναυδος με τις αλλαγές που έχουν γίνει στην πόλη μετά από τους αιώνες που πέρασαν. Ε, βλέποντα τα ρούχα που έχουν ε, βάλει άντρε και γυναίκε, αυτά που χρησιμοποιούνται πλέον, βλέποντα του υπολογιστέ, τα, τα κινητά, τι ε, τηλεοράσει, τα αυτοκίνητα, θα νόμιζε ότι έχει φτάσει σε ένα κόσμο δαιμονικό από τον 18ο αιώνα. Αν έρχονταν όμω στην ακρόαση ενό δικαστηρίου, την ακροαματική μάλλον διαδικασία ενό δικαστηρίου και απλώ παρίστατο στην εκδίκαση μια υπόθεση, θα καταλάβαινα ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στα δικαστήρια τη Ευρώπη και το εσωτερικό οικοδόμημα των δικαστηρίων, για να μην πω και ίδια τα έπιπλα των δικαστηρίων, οι πρωταγωνιστές του θεατρικού αυτού ε, έργου της δικαιοσύνης είναι το ίδιο. Οι ομιλίες και οι λόγοι είναι οι ίδιοι. Υπάρχει λοιπόν σαφής και επιτακτική ανάγκη να μεταρρυθμιστεί το δικαστικό σύστημα, η δικαιοσύνη, από το να προβλέπουμε εναλλακτικέ στο επίσημο δικαστικό σύστημα που, και στη δικαιοσύνη που παρέχουν τα κράτη. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται με αυτού που πιστεύουν ότι η διατησία έχει μέλλον, έχει πρόπτικέ, Όχι, εγώ νομίζω ότι η υποχρέωση των κρατών είναι να κάνουν μια βαθιά μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματο, όχι μόνο σε επίπεδο εκδίκαση και νομολογία, αλλά και πρακτικά στο τι συμβαίνει μέσα στα ίδια τα δικαστήρια. Είναι υποχρέωση του κράτου του δικαίου ε, να ε, καλύπτονται οι υποχρεώσει οι οικονομικέ και οι πολιτιστικέ και τις ίδιες τη δημοκρατία. Uh, Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Καλώ τον κύριο Ιβ Μπέχετς Βόγεμας, πρόεδρο της ομάδας εργασίας στο Συμβούλιο συμβολογράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θα ήθελε να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση του δικού του σχεδίου για τη διαμεσολάβηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχάς να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεσή της για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με ορισμένες πτυχές της διαμεσολάβησης σε θέματα αστικά και εμπορικά. Η διαπίστωση της κατάστασης είναι σαφής και εμφανίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνουμε ότι δεν, προβλέπει να αναθεωρήσει την οδηγία στο άμεσο μέλλον και το σκοπός της είναι να χρηματοδοτήσει έργα για τη διαμεσολάβηση μέσα από το πρόγραμμα ε, justice, δικαιοσύνη. Το Συμβούλιο Συμβολογράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφουγκράστηκε αυτό το κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεσμεύεται να πράξει τα δέοντα για να αναπτυχθεί η διαμεσολάβηση στην Ευρώπη. Σε πολλές χώρες τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα συμβολογράφο μπορεί να αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή με τον κοινοτικό του ρόλο, με το ρόλο του δημοσίου λειτουργού, του επικουρούντος στην δικαιοσύνη μεταξύ των ιδιωτών. Ο συμβολογράφο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση σε πολλά κράτη-μέλη. Έχει πολλαπλέ ε, αρμοδιότητε και στο δίκαιο κληρονομικό και στο εταιρικό και στο ε, δίκαιο το οικογενειακό. Είναι αυτός που εμπιστεύονται οι οικογένειες, αυτός που εμπιστεύονται οι επιχειρήσεις και γι' αυτό ο, ο συμβολογράφος θέτει στην υπηρεσία της διαμεσολάβησης τα ταλέντα και την εμπειρία του. Στο σχέδιο 2020, το Συμβούλιο Συμβολογράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβε τη δέσμευση να αναπτύξει τη διαμεσολάβηση στην Ευρώπη και γι' αυτό επιθυμούμε να δράξουμε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουμε πιο συγκεκριμένους στόχους. Να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο για την ε, πρακτική της διαβούλευσης στην Ευρώπη και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο Ευρωπαίων συμβολογράφων Παύλα Διαμεσολαβητών και έτσι να διευκολυθεί η συνεργασία του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δικτύωση συμβολογράφων διαμεσολαβητών στην Ευρώπη είναι προφανές ε, λόγω του ότι αυξάνονται εκθετικά οι φάκελοι σχετικοί και οι διασυνοριακές διαφορές, ε, τα θέματα που έχουν να κάνουν και με τις κληρονομιές άλλωστε. Και άρα η διευκόλυνση της συνεργασίας συμβολιογράφων μεταξύ ε, ε, διαφόρων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το θετικό και θα πρέπει να τεθούν εργαλεία στη διάθεσή τους και γι' αυτό εμείς αυτή τη στιγμή συγγράφουμε έναν οδηγό που θα λύσει θέματα ορολογίας ε, ρητρών που εφαρμόζονται ε, συνήθως μεταξύ άλλων. Οι Ευρωπαίοι συμβολεογράφοι έχουν επενδύσει πολλά στη διαμεσολάβηση εδώ και 10 χρόνια. Έχουν υπογραμμίσει τη δέσμευσή τους και δεσμεύονται να συνεχίσουν αυτές τις εργασίες επί τούτου και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό με το, έτσι ώστε να υπάρξει μια κοινή κουλτούρα για τη διαμεσολάβηση παγιωμένη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σα. Σας ευχαριστούμε κύριε Βάιντεμανς. Περνάμε στο δεύτερο μέρος του φωτοργαστηρίου και θα επικεντρωθούμε σε δύο πρακτικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα τα δυνατότητα να υπάρχουν συμφωνίες ε, διαιτησίας που να αναγνωρίζονται και να ε, επιβάλλονται ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση και έπειτα οι προκλήσεις της επιγραμμικής προσφοράς διαιτησίας. Θα προσκαλέσω τον καθηγητή Χωσέ Λουίς Ιγκλέσιας ε, από το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, έχει το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Με, ε, με τα δέκα λεπτά που μου επιτρέπει ο Πρόεδρος, μπορώ μόνο να σας κάνω μία σύνοψη όλων αυτών που έχουν σχέση με το ιδιωτικό δίκαιο και την διασυνοριακή επίλυση διαφορών για να καταλήξω σε μια σειρά μέτρων που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στους ευρωπαϊκούς κανόνες, στο ευρωπαϊκό δίκαιο για να βελτιωθεί αυτός ο τρόπος εξοδικαστικής επίλυσης διαφορών. Όλοι γνωρίζουν ότι η οδηγία του 2008 για τη διαμεσολάβηση περιορίζεται στη θέσπιση ενός ελάχιστου πλαισίου, νομικού πλαισίου ελάχιστου, ε, ε, έτσι, και έτσι δεν υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοί κανόνες συγκεκριμένοι του ιδιωτικού ε, διεθνούς δικαίου και αυτό δεν διευκολύνει τη μετακίνηση των πολιτών ούτε εξυπηρετούνται οι γενικότεροι σκοποί της οδηγίας με ομοιόμορφο τρόπο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαμεσολάβηση για τις συμβάσεις, καταρχήν Όλα αυτά διώπονται από, τα, από τον κανονισμό 1593 του 2008, Ρώμη 1. Επί της ουσίας όμως έχουμε ε, τους άλλους κανονισμούς που ισχύουν αναλόγως με το θέμα, το επίδικο. Για παράδειγμα, κανονισμός 650 του 2012, εάν η διαφορά έχει να κάνει με το mortis έχει να κάνει με διατροφικά θέματα η κανονισμο 4209 οταν εχει να κανει με διατροφικα θεματα για τη δικία και η διαφορά. Δηλαδή αλλάζει ο κανονισμός που ισχύει αναλόγως με την ουσία της υπόθεσης. Εφαρμόζονται όλα αυτά στη συμφωνία αναλόγως με το θέμα υπό τον όρο να, στη χώρα προέλευσης να είναι εκτελεστός ο συγκεκριμένος κανονισμός και να υπάρξει δημόσιο έγγραφο, αυτό είναι και το πιο συνηθισμένο, ή να υπάρξει και η πράξη δικαστική. Υπάρχουν δηλαδή αυτά τα εργαλεία, αλλά δεν καλύπτουν όλα τα αστικά και εμπορικά θέματα. Υπάρχουν μηχανισμοί εκτέλεσης διαφορετικοί και δεν είναι ενοποιημένη και νέα προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα που εγείρονται. Πέρα από αυτά τα εργαλεία έχουμε και τους εθνικούς κανόνες που θα πρέπει να ισχύσουν και να εφαρμοστούν. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα μοσαϊκό, δικαστικό και νομικό μοσαϊκό, πολύ κατακαιρματισμένο τοπίο με διαφορετικές συνθήκες και προϋποθέσεις που ισχύουν στα διάφορα κράτη-μέλη και άλλωστε δεν έχει λυθεί και το θέμα της διαμεσολάβησης ε, θέματα ιδιωτικών διαφορών. Έρχομαι στις επιλογές και στα μέτρα. Η διαμεσολάβηση γραπτή ε, καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις μεταρρυθμίσεων. Μία πρώτη επιλογή είναι αυτή που μας παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή να θεωρήσουμε ότι το υφιστάμενο σύστημα λειτουργεί εύλογα και λογικά, άρα δεν χρειάζεται να αναθεωρηθεί σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο η οδηγία. Αυτή είναι μια επιλογή. Α, επίσης, τα μέτρα που προτείνονται θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να εφαρμοστούν με εξα, εξατομικευμένο ή συνδυαστικό τρόπο και είναι ε, η εξή αυτή η επιλογή. Βεβαίως, να τροποποιηθεί το status quo γιατί τα στατιστικά στοιχεία και τα αποτελέσματα που έχουμε επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι σκοποί της οδηγίας. Άρα τα μέτρα βελτίωσης θα ήταν πια να αναθεωρηθεί πράγματι η εφιστάμενη οδηγία ή να εκπονηθεί νέο νομοθετικό εργαλείο. Είτε οδηγία είτε κανονισμός, όποιο και αν επιλέγει τελικά. Και θα πρέπει να δίδεται και να υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που θα καθορίζει το εφαρμοστέο δίκαιο όταν έχουμε διασυνοριακές διαφορές και να υπάρξει ε, αυτό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν τώρα υπάρχει σύγκρουση νομολογιών ή σύγκρουση ε, ε, νομοθεσιών και αν αυτό το εγχείρημα θεωρείται εξαιρετικά περίπλοκο ή προβληματικό, θα πρέπει το μέτρο να περιοριστεί μόνο σε επίπεδο εκτέλεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε διαφορετικό σημείο εστίασης. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια μεταρρύθμιση de Δηλαδή τους εκτελεστικούς και εφαρμοστικούς κανονισμούς να τροποποιήσουμε και να γίνει ρητή αναφορά στη Συμφωνία Διαμεσολάβησης και ρητός να αναφερθεί ότι το ισχυρό νομικό πλαίσιο είναι εφαρμοστέο μέσω των τρεγουσών συμφωνιών, κάτι το οποίο ισχύει και σήμερα, Είναι να συμπεριληφθεί ένα νέο κεφάλαιο για την αναγνώριση και εκτέλεση των συμφωνιών διαμεσολάβησης παράλληλα με τα κεφάλαια τα οποία ήδη υπάρχουν για τα δημόσια έγγραφα και τις ε, πράξεις δικαστικής ε, τις πράξει τη Θα μπορούσαμε να έχουμε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού διαμεσολάβησης και να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να εκπονηθεί αυτό το πιστοποιητικό διαμεσολάβησης και αυτό συνάδει με ήδη ισχύοντα νομικά εργαλεία, κανονισμός 850 του 2004 ή κανονισμός 650 του 2012 για το Μόρτις Κάουσα. Όλα αυτά ισχύουν σε όλα τα κρατημέλη χωρίς να υπάρξει καμία ειδική διαδικασία. Ε, άρα υπάρχουν παραλληλισμοί και θα μπορούσαμε αυτή την άγουσα να ακολουθήσουμε και στο ε, τομέα της διαμεσολάβησης. Μένει να διευκρινιστεί αν αυτό το πιστοποιητικό θα ήταν προαιρετικό ή υποχρεωτικό. Η προστιθέμενη αξία αυτού του πιστοποιητικού μου διαμεσολάβηση είναι η εξή. Θα υπάρχει ένα κοινό μοντέλο για την άμεση εφαρμογή και εκτέλεση των συμφωνιών και θα πρέπει ε, οι διαστάσεις που καλύπτονται να είναι πολύ πιο ευρείες από αυτές που καλύπτονται με τα υφιστάμενα εργαλεία οι επιφυλάξεις εικάζουμε ή έστω και αντίθεση ίσως ορισμένων κρατών μελών σε αυτή την επιλογή να συμπεριληφθούν οι ιδιωτικές συμφωνίες και τα ιδιωτικά συμφωνητικά είναι πράγματα που μπορούν να υπερπηδηθούν, να ξεπεραστούν αν έχουμε προαιρετικό σύστημα. Το έχουμε το προαιρετικό σύστημα στους άλλους κανονισμούς που σας ανέφερα. Άρα μπορούμε να έχουμε ένα διπλό σύστημα, ένα γενικό ε, και ε, μία δημόσια αρχή να έχει ε, μια δημόσια αρχή στη χώρα προέλευσης της συμφωνίας να έχει ε, πιστοποιήσει την αυθεντικότητα των αποφάσεων και να έχουμε και ένα προαιρετικό σύστημα για τα ιδιωτικά συμφωνητικά, τις ιδιωτικές συμφωνίες. Άλλη εναλλακτική επιλογή είναι η εξή να προβλέψουμε τουλάχιστον ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό διαμεσολάβησης περιορισμένου βεληνικού, περιορισμένης ισχύω για συγκεκριμένες διενέξεις ή για συγκεκριμένες κατηγορίες διάδικων μερών. Π.χ. διενέξεις μόνο για καταναλωτές, διαφορές μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσει. Βλέπετε ότι όλα αυτά τα ε, είδη ε, και όλες αυτές οι επιλογές ε, υπάρχουν και θα αξίζει να τις μελετήσουμε. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να τροποποιήσει το υφιστάμενο σύστημα και να εμπνευστεί από την αντίστοιχη Επιτροπή για το Εμπορικό Δίκαιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε εμπορικέ συμβάσει σε διεθνέ επίπεδο που θα προκύψουν από τη διαβούλευση που ε, λογικά θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2017. Οι αρχέ ε, αμυγό ιδιωτική φύση έχουν αναγνωριστεί και εκτελούνται οι αποφάσει αυτέ όταν τηρούνται ορισμένε προποθέσει. Και άλλωστε το κράτο κράτος που είναι ετών, που είναι ενάγων, έχει ε, άμυνα και δυνατότητες να προλάβει την εφαρμογή σύμφωνα με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958 για την αναγνώριση της εξτέλεσης των διαιτητικών αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση ε, όλα αυτά δεν είναι ξένα από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη και την Ένωμη Τάξη των κρατών μελών. Θα μπορούσαμε να εμπνευστούμε από τον νόμο 29 του 2013 το άρθρο 9 εδάφιο 4 της Πορτογαλίας, πορτογαλική νομοθεσία. Όταν μια συμφωνία διαμεσολάβησης έχει ε, γίνει σε άλλο κράτος μέλος και εκτελείται και εφαρμόζεται στην Πορτογαλία, άμεσα ε, γίνεται αυτό δεκτό και δεν χρειάζεται να αναγνωριστεί η συνάφεια με την πορτογαλική νομοθεσία. Δεν αντίκειται αυτό στην πορτογαλική ένωμη τάξη. Βλέπετε, μπορούμε να εμπνευστούμε λοιπόν από το πορτογαλικό δίκαιο. Μπορούμε να έχουμε τους απαραίτητους ελέγχους, τις ε, ασφαλιστικές δικλείδες και έτσι το ευρωπαϊκό μοντέλο εκτέλεσης των συμφωνιών διαμεσολάβησης μπορεί να μοιάζει με το υφιστάμενο που έχουμε για την αναγνώριση των συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε καλύτερη ομοιογένεια ε, Όλα αυτά θα ήταν ένα γρήγορο ε, και αποτελεσματικό εργαλείο για την επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει χρόνος για περισσότερες λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ καθηγητά για την άκρο ενδιαφέρουσα ε, ομιλία σας. Τελευταίος, αλλά εξίσου επιφανής, ο δόκτορας Γιν Χο από την Ολλανδία. Θα μας παρουσιάσει τις πρόσφατες εμπειρίες του με το μοναδικό σύστημα για την επίλυση διαφορών online το οποίο εφαρμόζεται ως πλατφόρμα στις ε, κατοχώρες ήδη. Έχετε 10 λεπτά κύριε Φερντόνσχο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ μέλη της Επιτροπής που με προσκαλέσατε στην ιδιότητά μου ως υπό την ιδιότητά μου ως ιδιότητα να σας παρουσιάσω αυτήν την πλατφόρμα για την επίλυση διαφορών που λειτουργεί ήδη στις κατοχώρες. Εδώ και δύο χρόνια με την υποστήριξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ολλανδίας και τον Δικηγορικό Σύλλογο της Ολλανδίας σχεδιάσαμε μία πλατφόρμα για τα διαζύγια. Είναι μια πλατφόρμα που βοηθάει τον κόσμο στις κάτω χώρες να χωρίσει. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο κόσμος αποτιμά τη διαδικασία διαζυγίου κατά 7,5% επιτυχή σε σχέση με τη χρήση της πλατφόρμας. Ε, δαπανούν λιγότερα ε, ευρώ από ό,τι στο παρελθόν για να, ε, λιγότερα χρήματα για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία γιατί τους παίρνει το πολύ πολύ τρεις μήνες η όλη διαδικασία. Κοιτάξαμε λοιπόν τα εργαλεία της διατησίας και τις διαδικασίες που επιτρέπει και επιτρέψαμε αυτό το κουτί εργαλείων να εκτυλιχθεί online. Ιδού κάποια από τα βασικά σημεία αφετηρίας. Νομίζω το καλύτερο είναι να σας δείξω λίγο την ίδια την πλατφόρμα για να καταλάβετε τι γίνεται. Και να σας πω ότι στις κάτω χώρες ο κόσμος μπορεί να πάει στον ιστότοπο. Είναι βεβαίως ε, Ολλανδική η βασική εκδοχή στις κάτω χώρες, αλλά έχουμε και άλλες γλώσσες. Είναι μια διαδικασία σε έξι στάδια, όπου επιτρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα μία διάγνωση για να δει κανείς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του. Μετά να δει τις προσδοκίες του, να περάσει σε ένα ερωτηματολόγιο βάσει των απαντήσεων του οποίου θα συγκεντρώσουμε εμεί νομικές πληροφορίες ανάλογα με την κατάσταση του καθενός και όταν αποφασίσει κανείς να προχωρήσει στο διαζύγιο μέσω αυτής της πλατφόρμας μπορεί online να ταυτοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική ταυτότητα ειδική από, την, από τις κυβερνητικούς φορείς με, μαγνητικά, με μαγνητικό τσιτ και να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τα παιδιά του, για μια σειρά από θέματα Όλα έχουν κατηγοριοποιηθεί σε πέντε κεφάλαια στην, ε, στο παράμερο της σελίδας και συγκεντρώνουμε πολλές ε, ερωτήσεις, έχουμε πολλές ερωτήσεις για το ποιες είναι οι ανάγκες του καθενός. Τι ανάγκες μπορεί να προκύπτουν σε σχέση με τα παιδιά. Μετά τους ζητάμε να μας πούν κάποιες από τις βασικές τους προσδοκίες ή ιδέες για το τι αποτελέσματα πιστεύουν θα πετύχουν μετά το διαζυγιό τους. Βασικά, Υπάρχει ε, μια σειρά λοιπόν από ερωτήσει στο ερωτηματολόγιο και όταν συγκεντρώσουμε τις απαντήσεις του πρώτου λαμβάνει μια ειδοποίηση το άλλο μέρος του διαζυγίου για να ειδοποιηθεί και να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Όταν και τα δύο μέρη έχουν συμπληρώσει τις ε, ερωτήσεις, έχουν δώσει τις απαντήσεις τους, περνούν σε ε, online διάλογο. Διευκολύνεται μέσω της πλατφόρμας η δυνατότητα να έχουν συζήτηση μεταξύ τους. Υπάρχουν εργαλεία διαλόγου στο κάτω μέρος της σελίδας και σε αυτό το μέρος της πλατφόρμας τους επιτρέπουμε με έναν ε, κορέκτορα να περάσουν σε online διάλογο, δηλαδή σε chat. Έχουμε αναπτύξει και κάποιους αλγόριθμους που επιτρέπουν το, στο σύστημα βάσει των αρχικών πληροφοριών και των δύο μερών ήδη να ετοιμάσει κάποια στελέχη κειμένου έτοιμα για να μπορέσουν ε, οι δύο πλευρές να περάσουν σε ένα βασικό κείμενο συμφωνίας. Έχουμε και πολλά εργαλεία υποστήριξη για να υπολογίσουμε λόγου χάρη πόσο θα κοστίσει η προστασία των παιδιών, η διατροφή. Εδώ βλέπουμε ότι χρειάζεται μια σειρά από συμφωνίε και ε, εμείς τα διευκολύνουμε όλα αυτά. Τα υποθάλπουμε. Υπάρχει λοιπόν μια φάση διαπραγμάτευση που να ολοκληρωθεί εδώ. Υπάρχουν πολλοί που χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη για να καταλήξουν σε συμφωνία. Αυτό που έχουμε συμπεριλάβει σε αυτή την πλατφόρμα είναι βασικά διαιτησία ε, βάση αιτήματο, on demand. Δηλαδή, όταν ε, πιστεύουν ότι έχουν κολλήσει στην επικοινωνία του οι πλευρέ ή ότι δεν μπορούν να τα πούν στον απέναντί του, δεν να τα πούν σε κάποιον εξωτερικό, φροντίζουμε να τους παρουσιάσουμε τρεις πιστοποιημένους και εκπαιδευμένους διαιτητές ακριβώς για αυτήν την online διαιτησία που διαθέτουμε. Έχουμε ειδικό πουλ με τέτοιους διαιτητές. Οπότε ένας θα μπει στη μέση και θα τους τα βρει. Θα περάσει σε συζήτηση μαζί τους αυτή την πλατφόρμα, με αυτές τις επιγραμμικές ε, διαιτησίες που μπορεί να πάρουν τη μορφή ενός τσάτ, ενός επιγραμμικού τσάτ των μερών με τον διαιτητή και μπορεί να αρχίσει να γίνεται συζήτηση. Και ξέρουμε ότι οι διαιτητές ε, ε, πολλές φορές προσφέρουν τη δυνατότητα να οργανωθεί και ζωντανά η διαιτησία γύρω από ένα τραπέζι, αλλά πολλές φορές έχουν το λάπτοπ μπροστά τους και με το λάπτοπ μπορούν να ανατρέξουν σε όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, συζητήσει φάσεις του διαλόγου που έχουν καταγραφεί στο σύστημα. Έτσι συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες, όλες οι συμφωνίες, όλες οι ανταλλαγές και επικοινωνίες ε, αποθηκεύονται και τηρούνται στα, στη μνήμη του συστήματος ώστε να χρησιμοποιηθούν όταν χρειαστεί. Επίσης υπάρχει και η κατοχήρωση, η απόδοση η απόφαση μάλλον κατόπιν αιτήματος. Δηλαδή κάποιος τους βοηθά ουσιαστικά, ο διαιτητή, να καταλήξουν σε μια απόφαση. Κατοχυρώνεται η απόφαση στην πλατφόρμα. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιείται μια κραματική διαδικασία, όπως λέγεται, με τα online εργαλεία που σας εξήγησα, με τον ίδιο περίπου τρόπο. Και τι γίνεται με αυτό. Αυτό δίνει την εγγύηση ότι οι πλευρέ που θα επιλέξουν αυτή την πλατφόρμα μπορούν πραγματικά να ολοκληρώσουν το διαζύγιο του, να χωρίσουν εντελώ. Μπορεί να χρειάζεται επιπλέον προστασία βεβαίω και κάποια χέγγυα, όπω είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ. Χρειάζεται λοιπόν μια ουδέτερη επισκόπηση στο τέλο και εκεί έρχεται και μπαίνει στη μέση ένα ειδικό δικηγόρο οικογενειακού δικαίου, ο οποίο αποτιμά την αμεροληψία, την ουδετερότητα, την πλήρη συνένεση στο διαζύγιο, το γεγονό ότι οι πλευρέ του αδυναμότερου μέρου έχουν προστατευθεί και ότι δεν αναγκάζεται, δεν εκβιάζεται να δώσει κάτι που δεν θέλει το άλλο μέρο. Έτσι, έχουμε επιτρέψει 5% των διαζυγίων στις κάτω χώρες τους τελευταίους 18 μήνες να περάσουν από αυτή την πλατφόρμα. Δηλαδή περίπου 350 άνθρωποι έχουν χωρίσει έτσι. Απλώς να πω ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ε, οι διαζευγμένοι έχουν αποτιμήσει την όλη εμπειρία του διαζυγίου με 7,5 στα 10. Οπότε ε, έχουμε κάνει πρόσφατα, ξεκινήσει μάλλον πρόσφατα μια μελέτη ικανοποίηση μετά το διαζύγιο και έξι μήνες ε, μετά οι ίδιοι που είχαν απαντήσει θετικά συνεχίζουν να δίνουν βαθμό 7,5 στο διαζύγιό τους. Αλλά μετά την ελλαγή αυτή ε, οι διαζευμένοι μπορεί να δουν ότι οι συμφωνίε τι οποίε κατέληξαν στην όλη πλατφόρμα και στην όλη διαδικασία τη δεν είναι οι καλύτερε. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα συστηματικά, ένα τρίμηνο, ένα εξάμηνο, ένα χρόνο, αν θέλουμε, να πηγαίνουμε πάλι στην πλατφόρμα για να προσαρμόζουμε τη συμφωνία. Αν προκύψουν νέε διαφορέ για οτιδήποτε. Για την ε, προστασία των παιδιών, για την κυδαιμονία, για τα λεφτά, τη διατροφή. Μπορεί να πάει κανεί στην πλατφόρμα και με τα ίδια εργαλεία υποστήριξη, με του ίδιου επαγγελματίε, ε, μπορούν να βρουν πάλι λύσεις online. Αυτό το είδος οι πλατφόρμες, αυτές οι κοινοτόμες λύσεις ουσιαστικά αλλάζουν, αλλάζουν την αντίληψη που έχουμε για τη διαδικασία της διευθυνσία πλέον. Ακόμη και την ε, ιδέα που έχουμε σχηματίσει στα κεφάλια μας για την ακροαματική διαδικασία στα δικαστήρια. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες βεβαίω στην πράξη, διότι βλέπουμε ότι παραδοσιακά οι κανόνες που διευθετούν τους το πώς εργάζονται οι επαγγελματίες, οι δικηγόροι και οι διαιτητέ, δεν ε, συνδυάζονται με τι ανάγκε αυτού του συστήματος. Λόγω χάρη στι κατοχώρε, η νομοθεσία για τους δικηγόρου και του διαιτητέ απαιτούν να έχουν πρόσωπο με πρόσωπο επαφή και ο καθένα να εμφανίζει το διαβατήριό του κάθε φορά που οργανώνεται συνάντηση. Εδώ έχουμε ε, χρησιμοποιήσει, όπω σα είπα, το μηχανισμό ταυτοποίηση ε, που έχει τη σφραγίδα τη κυβέρνηση, που βάσει των κανόνων αυτών δεν θα ήταν εφεμητό ούτε νόμιμο, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί για φορολογικού σκοπού και για κάθε επικοινωνία με την κυβέρνηση είναι έγκυρο. Νομίζω λοιπόν ένα από τα πράγματα που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι Πρέπει να δούμε πώς θα ενθαρρύνουμε αυτού του είδους την διευθέτηση. Πώς μπορούμε να εξυγχρονίσουμε και να καινοτομήσουμε να επιτρέψουμε να χρησιμοποιούνται περισσότερο τέτοιε καινοτόμε λύσει και ίσω να αφήσουμε λίγο περισσότερο χώρο για πανεστατικές λύσει. Λίγη ελευθερία για αυτό το περιβάλλον το νομικό. Να δούμε οι πολίτε τι θέλουν. Είναι κάτι το απαραίτητο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φερντός για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα ε, παρουσίαση. Να ξεκινήσουμε τώρα το δεύτερο γύρο ε, ερωτήσεων και απαντήσεων με τους ε, προσκεκλημένους μας. Θα ήθελα να καλέσω τόσο τα μέλη αλλά και τα μη μέλη αυτή τη στιγμή να θέσουν τα ερωτήματά τους εφόσον το επιθυμούν αλλά με έναν χρονικό ορίζοντα 10 λεπτών. Πολύ αυστηρό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές εκ μέρους της Κομισιόν για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις. Όσον αφορά την παρουσίαση, την πολύ ενδιαφέρουσα ε, παρουσίαση του καθηγητή Ιγκλέσιας, θα ήθελα να αναφέρω ότι η Κομισιόν, ε, βάσει και του θεσμικού της ρόλου, και σε στενό συντονισμό με τα κράτη-μέλη, εκπροσωπεί την Ένωση στις ε, διαπραγματεύσεις Γιούν Σιτράλ, ε, ένας μηχανισμού που αφορά την ε, διεθνή επίλυση διαφορών. Και θα ήθελα στο πλαίσιο αυτό να αναφέρω ότι Ανάλογα με την τελική μορφή του Σιτραλ και το περιεχόμενο του εργαλείου αυτού, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να ε, ενταχθεί σε αυτόν τον μηχανισμό, αυτός ο μηχανισμός προφανώς δεν ε, θα αφορά μόνο την ε, επίλυση διαφορών εκτός Ένωσης, αλλά και εντός Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Professor Iglesias, would you like to respond to... Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο αυτό είναι υπό συζήτηση ακόμα. Ε, η διαπραγμάτευση γίνεται για τον ορισμό που είναι εξαιρετικά ευρύς. Και βεβαίως εκεί θα περιληφθεί και η σημερινή μορφή της, δια, της διατησίας, διαμεσολάβησης, με Και όπως είπα στην, στην πολύ σύντομη και γρήγορη παρουσίασή μου, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει αυτή τη συμφωνία και έχει την ιδιοκτησία αυτής, λόγω αρμοδιοτήτων που έχει και για εξωτερικά θέματα, τότε βεβαίως και θα είχαμε διαμεσολάβηση εφαρμόσιμη και εφαρμοστέα στις ενδοκοινοτικές υποθέσεις και αυτή η διαμεσολάβηση θα είναι παρεμφερής και ταυτόσιμη με αυτήν που ισχύει και εφαρμόζεται εντός και εκτός Ευρώπης για τις συμφωνίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα τρίτα μέρη, με τρίτα κράτη, όπως σας είπα στην παρουσίασή μου. Υπ' αυτή την έννοια μου φαίνεται εξαιρετικά καλό όλο αυτό και ελπίζω αυτή η διαπραγμάτευση να φτάσει σε αίσιο τέλος, να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτή την εκπεφρασμένη βούληση να δράσει σε αυτό το τομέα εξ ονόματος της Ένωσης. Thank you, professor. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Ο κύριος μου. έχει ζητήσει το λόγο για να θέσει ένα ερώτημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές για την παρουσία τους, για τα επιχειρήματά τους, τις παρουσιάσεις τους, εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματι. Δύο ερωτήματα έχω να θέσω. Πρώτον, ως προς την πρόταση δημιουργίας Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Διαμεσολάβησης. Είναι μια πρόταση η οποία με εκπλήσει κάπως, γιατί κατανοώ από τη μία την ανάγκη να καταρτιστεί σωστά ο διαμεσολαβητής, όμως τα κράτη θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτό το μέλημα και να τα ενθαρρύνουμε κιόλας σε αυτό το εγχείρημα κατάρτισης. Νομίζω ότι έτσι στρεβλώνουμε την αρχή της επικουρικότητας ή της θέτουμε εμπόδια σε κάθε περίπτωση. Δεύτερον, για το διαδικτυακό διαζύγιο στις κάτω χώρες. Μαθαίνω ότι λειτουργεί πολύ καλά. Αυτό το οποίο με εκπλήσει είναι το εξής. Από μόνο του ένα διαζύγιο είναι απλό. Ε, λιγότερο απλό είναι ο αντίκτυπος τα αγαθά και στην περιουσία τα οποία θα πρέπει να μοιραστούν. Και υπάρχει και πρόβλημα με την επιμελητία, με την κυδαιμονία των παιδιών. Αυτά τα προβλήματα ε, έχουν απόσταση από το διαζύγιο αυτό κάθε αυτό και εκεί σε αυτά τα προβλήματα δεν φτάνει ούτε η διαμεσολάβηση ούτε το διαδικτυακό διαζύγιο. Πολύ συχνά είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε στο δικαστήριο για την επίλυση αυτών των θεμάτων. Και αυτές είναι οι δύο μου ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ωραία, θα ήθελαν οι ομιλητές μας να τοποθετηθούν. Eh, ναι, σε ό,τι αφορά ε, στο πρώτο ερώτημα, το προτινόμενο πιστοποιητικό διαμεσολάβηση στην Ευρώπη, ίσως δεν έγινε απολύτως αντιληπτό. Αυτό το οποίο εγώ ήθελα να πω είναι το εξής. Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Διαμεσολάβησης δεν θα έχει καμία σχέση με το διαμεσολαβητή. Θα είναι ένα πιστοποιητικό το οποίο θα εκδίδεται άπαξ μόλις έχει υπάρξει συμφωνία διαμεσολάβησης, έχουν φτάσει τα μέρη τα διάδικα σε αυτή τη συμφωνία, είναι εκτελεστό και θα πρέπει να εκτελεστεί η συμφωνία αυτή σε άλλη χώρα μέλος διαφορετική από τη χώρα προέλευσης. Το ίδιο γίνεται και με το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Κληρονομιών το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Διαμεσολάβησης θα διαδραματίσει επακριβώς τον ίδιο ρόλο. Δηλαδή θα χρησιμεύει, το προτείνουμε, για να χρησιμεύσει, για να αποφευχθεί όλη αυτή η διαδικασία παρόλο που έχει απλουστευτεί του εξεκβάτουρ, δηλαδή της εκτέλεσης του να κηρυχθεί εκτελεστός ο τίτλος του ε, της δικαστικής απόφασης που έχει βγει στο άλλο κράτος μέλος. Αυτός είναι ο σκοπός που εξυπηρετεί. Ότι δηλαδή η δημόσια αρχή της εκάστοτε χώρας έχει επιστοποιήσει το εξεκβάτουρ, το εκτελεστέο της απόφασης σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Επομένως αυτό προτείνουμε να ισχύσει και για το πιστοποιητικό διαμεσολάβησης. Τώρα, θα πρέπει να μελετηθεί αυτό που λέτε, είναι άλλο θέμα. Θα μπορούσαμε ίσως να ακολουθήσουμε τη γραμμή των εργασιών που γίνονται στην αντίστοιχη Επιτροπή του Οργανισμού Εθνών για την επίλυση των εμπορικών διαφορών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα, γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβω ότι δεν ήμουν επαρκώς σαφής. Να σας πω δηλαδή ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτήν την πλατφόρμα στο τέλος έχουν διαζύγιο που αφορά και συμπεριλαμβάνει την, τον διαμορισμό των περισσότερων στοιχείων, τις κατοικίες τους, όλες οι διευθετήσεις που σχετίζονται με τα παιδιά, την κυδαιμονία, τη λήψη από κοινού αποφάσεων, την διατροφή ε, για τα παιδιά και για τον πρώην σύζυγο. Απλά το θέμα είναι ότι μέσω μιας τέτοιας κεντρικής πλατφόρμας μπορούμε να εντάξουμε ε, και την οικονομική εμπειρογνωμοσύνη οικονομικών πτυχών. Όταν για παράδειγμα πρέπει κανείς να εκτιμήσει την αξία μιας κατοικίας, του σπιτιού του, ε, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες διευθετήσεις ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα όλων των μέρων με τρόπο που θα αντικατοπτρίζει και αυτήν την ενημερωμένη συγκατάθεση. Για να το θέσω πολύ απλά, ε, στην ουσία με το κλικ ενός κουμπιού έχει κανείς πρόσβαση σε εμπειρογνώμονα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν εντάσσουμε την υποστήριξη που ε, ε, χρειάζονται οι ε, ε, άνθρωποι που παίρνουν το διαζύγιο. Όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ε, αντιμετωπίζουμε βεβαίως ε, τις δυσκολίες ε, της μετάβασης από τη μία διαδικασία στην άλλη διαδικασία. Στο τέλος δηλαδή, προφανώς οι άνθρωποι ε, πρέπει να στείλουν τη συμφωνία τους σε δικαστή, γιατί δικαστής πρέπει να εγκρίνει ε, την έντυπη μορφή αυτής της συμφωνίας και κατά μέσο όρο αυτή η διαδικασία διαρκεί τρεις μήνες. Τρεις μήνες ε, και στη συνέχεια απαιτούνται άλλες τέσσερις εβδομάδες έως την έγκριση από το δικαστήριο. Κάτι αυτό, για παράδειγμα, μπορεί να βελτιωθεί αν ε, καταφέρουμε να καταστήσουμε την μετάβαση από τη μία διαδικασία στην άλλη ομαλότερη. Για ένα λεπτό, κύριε καθηγητά. Θέλω να μιλήσω στους δύο ευρωβουλευτές, ε, γιατί ρώτησαν τι είναι η διαιτησία. Το ερώτημα ε, αφενός ήταν γιατί θα πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι αξίζει να ε, χρηματοδοτηθεί η διαμεσολάβηση, γιατί δεν βελτιώνουμε απλά την, ε, τα δικαστήρια. Γιατί, ρωτήσατε εσείς, γιατί να προωθήσουμε τη διαμεσολάβηση εφόσον οι υποθέσεις στις περισσότερες κατά καταλήγουν στα δικαστήρια. Εδώ μιλάμε για την πεμπτουσία του ζητήματος. Εδώ δεν είναι διαζευτικό είτε διαμεσολάβηση είτε δικαστήρια. Το ζητούμενο είναι οι άνθρωποι να έχουν στη διάθεσή τους μια διαφορετική επιλογή. Αναφερθήκατε για παράδειγμα στο ζήτημα του χρόνου και του κόστους. Αλλά αυτό είναι μόνο μία πτυχή του ζητήματος. Δεν μπορούμε να έχουμε δικαστήρια τα οποία να τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι ε, εφικτό. Η διαμεσολάβηση, η διατησία είναι πολύ πιο γρήγορη. Αυτό όμως αφορά το ποσοτικό κομμάτι. Υπάρχει και ένα ποιοτικό. Τι είδους συμφωνία μπορεί κανείς να ε, ε, πάρει στα χέρια του. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης έχουμε περίπου 25 εκατομμύρια αστικές υποθέσεις αυτή το 2016. Ας πούμε ότι βρίσκονται 50 εκατομμύρια άνθρωποι ενώπιον των δικαστηρίων. Τι γνωρίζουμε για αυτούς τους 50 εκατομμύρια ανθρώπους ένα πράγμα. Και μόνο. Ότι 25 ε, ε, εκατομμύρια αυτών των ανθρώπων δεν θα δικαιωθούν. Δεν θα πάρουν αυτό που θέλουν, θα πρέπει να πληρώσουν. Μήπως εκ των προτέρων θα μπορούσαν να ενημερωθούν ότι υπάρχει και μια εναλλακτική μορφή συμφωνίας. Ε, σκεφτείτε και κάτι άλλο. Ε, ή άκουσα ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο το 3% των υποθέσεων που ξεκινούν στα δικαστήρια τελικά ε, καταλήγουν σε πλήρη δικαστική διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι 97% των περιπτώσεων ε, ε, καταλήγουν σε συμβιβασμό εξοδικαστικό. Μήπως θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε αυτή τη διαδικασία μέσω ευαισθητοποίησης, μέσω της υποστήριξης. Αυτό είναι και η ουσία. Η διαιτησία αφορά και τα δύο πράγματα. Κάνουμε διαμεσολάβηση, βελτιώνουμε και τα δικαστήρια είναι, κάτι που μπορεί να, είναι δύο πράγματα που μπορούν να συνεπάρξουν και ταυτόχρονα ε, ε διευρύνουμε την γάμα των επιλογών για τους πολίτες. Αυτό είναι το βασικό. Και δεύτερον, ε, το ζήτημα αυτό αφορά και τον υποχρεωτικό ή τον ε, εθελοντικό δικαστικό της, της διαμεσολάβησης. Δεν χρειάζεται να είναι είτε το ένα είτε το άλλο. Μπορεί να, μπορεί να απαιτούνται διάφορα βήματα ώστε να παροτρινθούν τα διάδικα μέρη να ακολουθήσουν τη διαμεσολάβηση. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει για να βελτιώσουμε όλοι το έργο μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στέφεκ για 30 δευτερόλεπτα γιατί μας τελειώνει ο χρόνος. Πολύ σύντομα. Θέλω να απαντήσω σε αυτά που ακούστηκαν. Η διαμεσολάβηση και τα δικαστήρια δεν αφορούν μόνο τα χρήματα και τον χρόνο. Αφορούν τα συμφέροντα των ίδιων των πολιτών. Και αν διαβάσουμε ε, με σοβαρότητα την, θεμελιο, την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή επικεντρώνει στους πολίτες. Και ποιος ξέρει καλύτερα ποια είναι η καλύτερη λύση. Είναι το κράτος ή ο πολίτης, μέσω, το κράτος μέσω των ε, νόμων και των δικαστήριων. Εγώ θα έλεγα ότι η απάντηση είναι ότι ε, οι πολίτες γνωρίζουν καλύτερα τα συμβαίροντά τους από οποιονδήποτε άλλο. Οπότε μπορούμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τέτοια μέσα, φυσικά βεβαίω, γιατί να μην το κάνουμε, φυσικά τα δικαστήρια αποτελούν την έσχατη λύση. Αν οι πολίτες της Γαλλικής Επανάστασης ε, έρχονταν σήμερα στις Βρυξέλλες, θα ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι με τη διαμεσολάβηση. Γιατί, γιατί η Επανάσταση, η Γαλλική Επανάσταση αφορούσε τη δημοκρατία, η οποία δίνει την εξουσία στον λαό. Αν λοιπόν ε, η επίλυση διαφορών ε, είναι κάτι που πρέπει να θέλουμε να το δώσουμε ε, στους πολίτες. Ε, αυτό ε, είναι μια λύση για το μέλλον. Αλλά 30... Ο κύριος Μαρίνιο Επίλτο. Ευχαριστώ. Όμως το ζήτημα είναι ότι η διαιτησία δεν μπορεί να είναι εναλλακτική στα επίσημα δικαστήρια. Τα δικαστήρια έχουν ε, ειδική ε, περίπτωση συνδιαλλαγής ε, για να βρεθεί μια λύση εξοδικαστική. Εδώ μιλάμε για κάτι εκτός δικαστικού συστήματος που ουσιαστικά εκμεταλλεύονται το αρνητικό στοιχείο που μπορεί να έχουν τα δικαστήρια και μία απάντηση, παρατήρηση μάλλον για την πλατφόρμα για τα διαζύγια και τη θέση που μπορεί να έχει εδώ το δικαστήριο. Όσοι έχουν υπογράψει εδώ την ε, συμφωνία έχουν μιλήσει ενώπιον δικαστή. Ο δικαστής πριν αποδώσει μια απόφαση γνωρίζει επαρακριβώς εάν τα μέρη ε, γνωρίζουν τι ε, επιφέρει η συμφωνία την οποία υπογράφουν. Τι κερδίζει και τι χάνει ο καθένα. Αυτό ακριβώ είναι το κέρδο των δικαστηρίων. Και εκεί είναι και το πρόβλημα. Να μην γνωρίζουν τα μέρη πώ θα προστατεύσουν ακριβώ τα δικαιώματά του. Διότι η γλώσσα του δικαστηρίου δεν είναι πάντοτε ε, προσβάσιμη σε όλου του πολίτε. Ο δικαστή, ο οποίο απλώ περιορίζεται στο να ε, αποδώσει μια γραπτή απόφαση, πολλέ φορέ μπορεί να έχει γίνει χωρίς να γνωρίζουν τα μέρη ε, ακριβώς τι συμβαίνει, ιδίω το πλέον ε, οικονομικά δύναμο μέρος. Άρα δεν μπορεί κανείς να παρακάμπτει τα δικαστήρια Εδώ το να χαλάμε χρήμα για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημα, που δεν ξέρουν τι θα πει αντίφαση, αντιπαραβολή, όλοι αυτοί οι κανόνες που κάνουν το δικαστικό σύστημα να λειτουργεί, μπορεί τελικά να ζημιώνει τα μέρη και να είναι και εξαπάτηση της ίδιας της δικαιοσύνης. So, thank you so much. Ωραία, ευχαριστώ. Λόρδε Φως, για 20 δευτερόλεπτα παρακαλώ. Δύο σημεία. Απαντώντας στον ε, Πορτογάλο Ευρωβουλευτή. Η απάντηση είναι τα δικαστήρια πρέπει να είναι πιο γρήγορα και λιγότερο δαπανηρά. Αυτό είναι στόχος για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κάνουμε, ακούσατε και από τον Ολλανδό συνάδελφο, ότι πατάς κουμπί και ε, λαμβάνεται απόφαση. Δεν μπορεί, να κάνεις, δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα πιο γρήγορα από αυτό. Δεύτερο σημείο, η διαμεσολάβηση διαφέρει από την εκδίκαση μιας υπόθεσης, διότι η διαμεσολάβηση προσφέρει λύση την οποία αποδέχονται και τα δύο μέρη και γι' αυτόν τον λόγο είναι περισσότερο ικανοποιημένα, ακριβώς γιατί έχουν αποδεχθεί μία ε, λύση, ενώ στην εκδίκαση ε, το ένα μέρος ε, δεν είναι, πάντοτε ε, μέρος που δεν, έχει, δεν έχουν ικανοποιηθεί τα δικά του αιτήματα. Λοιπόν, με την ιδιότητα του εισηγητή για την έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία για τη διαμεσολάβηση θα προσπαθήσω να εξάγω κάποια συμπεράσματα. Όπως είπε ο κύριος Χάιμπαχ, η εφαρμογή της οδηγίας για τη μεσολάβηση είχε σημαντικότατη επίπτωση στην ομοθεσία πολλών κρατών μελών πέραν της θέσπισης ορισμένων απαιτήσεων για τις διασυνοριακές αποθέσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, είναι ε, σημαντικό να σημειωθεί ότι η οδηγία οδήγησε στη διεύρυνση της χρήσης της διαμεσολάβησης και σε εγχώριες ε, υποθέσεις, καθώς τα περισσότερα κράτη-μέλη διεύρυναν ε, την, ε, το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία και πλέον καλύπτονται και οι εγχώριες, ε, οι, υποθέσεις. Έτσι λοιπόν η οδηγία έχει προστιθόμενη ευρωπαϊκή αξία. Αφετέρου όμως οι δυσκολίες που σχετίζονται με τα συστήματα λειτουργίας της διαμεσολάβησης ε, σχετίζονται με την διαφορετική κουλτούρα που επικρατεί στις περισσότερες χώρες καθώς και στην ε, περιορισμένη ευαισθητοποίηση ε, γύρω από την διαμεσολάβηση και την κακή λειτουργία των μηχανισμών εξασφάλισης ποιότητας οι περισσότερες, στις περισσότερες περιπτώσεις οι πολίτες δεν αξιοποιούν στο βαθμό που, θα ήταν επιθεμητό την διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση χρησιμοποιείται σπάνια συστηματικά από διάδικα μέρη και από δικηγόρους. Όσον αφορά τη διαδικασία για την επίτευξη μιας ισορροπημένης σχέσης μεταξύ διαιτησίας και δικαστικών, δικαστικών διαδικασιών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία για τη διαμεσολάβηση επιδιώκει να ενθαρρύνει περισσότερους πολίτες να χρησιμοποιήσουν τη διαμεσολάβηση και να εξασφαλίσει μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ διατησίας και δικαστηρίων. Ωστόσο, οχτώ χρόνια μετά την υιοθέτηση αυτής της οδηγίας, φαίνεται ότι οι θεμελιώδεις στόχοι της δεν έχουν ακόμη ε, επιτευχθεί. Η διαμεσολάβηση χρησιμοποιείται σε λιγότερο από το 1% των υποθέσεων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνη η εξαίρεση ε, είναι το μοντέλο ε, αρχικής διαμεσολάβησης που χρησιμοποιείται στην Ιταλία, όπου 81% όλων των αστικών υποθέσεων πρέπει πρώτα να περάσουν από μια αρχική τουλάχιστον φάση ε, διαμεσολάβησης. Αυτό αναδεικνύεται ως βέλτιστη πρακτική. Στις συνθήκες αυτές προτείνεται ο Ευρωπαίος Νομοθέτης να ε, αναθεωρήσει το άρθρο 5 της οδηγίας ε, ώστε να απαιτείται από τα, ε, από διάδικα μέρη να συμμετέχουν σε μια αρχική τουλάχιστον φάση διαμεσολάβησης με εκπαιδευμένο διαμεσολαβητή. Θα είναι μια διαδικασία ταχεία και όχι δαπανηρή. Πρέπει να τονιστεί ότι η ισορροπημένη σχέση μεταξύ διαμεσολάβησης και δικαστηριών θα μπορούσε να εξοικονομήσει εκατομμύρια ευρώ και εκατομμύρια ε, περιττών ημερών εκδίκασης υποθέσεων στα δικαστήρια. Η διαμεσολάβηση λοιπόν έχει πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο το 22% των συνολικών ε, ε, ανέρχεται μόνο στο 22% των συνολικών ε, κόστων του ε, δικαστικού συστήματος. Όπως είπε και ο Lord Justice στην παρουσίασή του, δημιουργήθηκε ένα κοινό έργο το, στις αρχές του 2016 μεταξύ του ε, Ευρωπαϊκού Δικτύου Συμβούλων για τη Δικαστική Εξουσία και των Συμβουλιογράφων. Το, το έργο αυτό έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου ε, για τις διάφορες μορφές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Σκοπός είναι να υπάρξει διαβούλευση και να ε, συνταχθεί ένα έγγραφο στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι απόψεις των Ευρωπαίων εμπλεκόμενων φορέων. Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της διατησίας και άλλων μορφών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως παρουσίασε ο κ. Στέφεκ, πρέπει να αναφερθεί ότι η εις ανάλυση των ζητημάτων αυτών, η οδηγία για τη διαμεσολάβηση, οι οδηγίες ADR και ODR έχουν επιτύχει ορισμένες βελτιώσεις στο θέμα αυτό, αλλά ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικότατες ελλείψεις. Το νομικό τοπίο ε, των δυνατοτήτων εναλλακτική επίλυση διαφορών είναι ακόμη ασαφέ. Η οδηγία για τη μεσολάβηση αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό εργαλείο που ε, αφορά συγκεκριμένη μορφή εναλλακτική επιλύσης διαφορών. Η οδηγία EDR και ο κανονισμός ODR ε, υιοθετούν μια γενική μόνο προσέγγιση όσον αφορά την εναλλακτική επέλυση διαφορών και δεν διακρίνουν μεταξύ των διαφόρων μορφών εναλλακτική επίλυση διαφορών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Επιπλέον, αυτά τα εργαλεία ορόσημα αφορούν κυρίως τη σχέση μεταξύ της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και των δικαστικών διαδικασιών και αφορούν ε, τις, ε, και, λιγότερο τις ε, συγκεκριμένες μορφές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Η απουσία μια βασική αρχή, όσον αφορά τη ρύθμιση τη εναλλακτική επίλυση διαφορών είναι ο κυριότερος λόγο για τις ελλείψει τη χρήση αυτών των εναλλακτικών μορφών επίλυση διαφορών για του πολίτε. Οι νόμοι στον τομέα αυτών είναι κατακαιρματισμένοι και ανεπαρκεί και ω εκ τούτου οι πολίτε δεν επιλέγουν τη μορφή εναλλακτική επίλυση διαφορών που αντιστοιχεί καλύτερα στα δικά τους ε, συμφέροντα. Τρει λύσει. Ε, προτείνονται ε, ε, εργαλεία για την επίλυση διαφορών, δίκτυα για τη συνεργασία και τρίτον ένα πλαίσιο για την θέσπιση των αρχών που θα διέπουν την επίλυση διαφορών. Όσον αφορά σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ διατησία ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, υπάρχουν θέματα που εγείρονται για τη διασυνοριακή διατησία και ο καθηγητής Ιγκλέσιας είπε ότι η υπόθεση αυτή τον έχει, αφορέ, τον τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και είναι και άμεσα σχετισμένη με την ενοποίηση της Ευρώπης. Η ενεργοποίηση της οδηγίας περί έχει να κάνει με την παρουσία της και την εφαρμογή της οδηγίας αυτής στα κάτι μελη Όμως είναι πολλές οι σημαντικές διαφορές, όπως η απουσία ε, ιδιωτικών κανόνων και διασυνοριακών συμφωνιών. Οπότε είναι θέμα το τι νομικό πλαίσιο δημιουργείται για να ε, είναι σαφείς οι βασικές αρχές της διατησίας. Όπως είπε ο καθηγητής Ιγκλέσιας, για να μπορέσουν οι πολίτες να εμπιστευτούν πλήρως το σύστημα διατησίας στο μέλλον, τουλάχιστον ό,τι αφορά τη διασυνοριακή επίλυση διαφορών, πρέπει να υπάρξει πλήρης κυκλοφορία, ανεμπόδιστη κυκλοφορία όλων των σχετικών κανόνων σε κάθε κάτος μέλος και κάθε κάτος μέλος θα πρέπει να είναι ασφαλές ε, για το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ένωση. Έτσι θα έχουμε ε, κάποιους βασικούς κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου για βασικές πτυχές της διετησίας, αλλά έτσι και φτηνούς, απλούς τρόπους για την επιβολή των διασυνοριακών συμφωνιών ανά την Ένωση σε ό,τι αφορά τις νομικές και πρακτικές ε, επιπλοκές της επιγραμμικής διαιτησίας, ιδίως την online διαιτησία και επίλυση διαφορών, οι πλατφόρμες ε, που προτάθηκαν στις κάτω χώρες είναι μια καινοτόμως λύση για τις υπάρχουσες διαδικασίες σε ένα επιγραμμικό περιβάλλον. διότι το τωρινό σύστημα θα μπορούσε να βελτιωθεί. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες δυσκολίες που δεν επιτρέπουν να φτάσει το πλήρες δυναμικό της σε πλατφόρμα για τους πολίτες. Οι πολιτικοί ηθήνοντες πρέπει να διευκολύνουν και να τονώσουν την περαιτέρω πρόοδο της επιγραμμικής online επίλυση διαφορών. Μια σημαντική πτυχή θα μπορούσε να είναι να δημιουργηθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει και τονώνει περισσότερες ε, πειραματικές ε, τέτοιες προσπάθειες, ώστε οι επιγραμμικές καινοτόμες λύσεις να δοκιμάζονται στην πράξη σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σε μικρή κλίμακα, ώστε ο αντίκτυπός τους να αξιολογείται γρήγορα. Οι εξελίξεις αυτές επιτρέπουν τα δικαστήρια να ε, επιβάλλουν τις αποφάσεις τους ε, εφόσον χρειαστεί και δεν λειτουργήσουν οι πλατφόρμες διετησίας. Είναι σημαντικό αυτό από την ε, μακροκαθημερινότητα και την μακροσκοπική διάσταση των πραγμάτων. Εφόσον υπάρξουν αυτέ οι εφαρμογέ των δικαστηρίων, θα υπάρχει περισσότερη ευελιξία για τον νομοθέτη και τον πολιτικό ηθήνοντα σε σχέση με τη διατησία και προκειμένου να αντιμετωπίσει το ένα και πιο περίπλοκο δίκτυο απαιτήσεων που έχουν δημιουργηθεί από την παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστούμε πολύ. Και ας ελπίσουμε να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση για την υλοποίηση της οδηγίας περί